because good morning. Good morning, colleagues. Can we settle down? Καθίστε παρακαλώ, προσδεθείτε, μην καπνίζετε. Welcome to transport colleagues and... Χαιρετίζω τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και όλους αυτούς που δεν είναι κανονικά παρόντες στις συνεδριάσεις μας της Επιτροπής Μεταφορών τους Καλωσορίζω όλους συλλήβδην και περνώ στις ε, ανακοινώσεις μετά από τις συνεδριάσεις των συντονιστών, αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση των συντονιστών. Προηγουμένως να σας πω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας, αλλά η αίθουσα αυτή είναι κάπως διαφορετική έχει μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητος από ό,τι έχουμε συνήθως και ενώ διαβιβάζεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας δεν θα έχουμε τις ε, φυσιολογικές ε, δυνατότητες για να φαίνεται το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών κτλ. Αλλά για αυτούς που έρχονται στην αίθουσα μόλις, ζητώ συγγνώμη, αλλά παρόλα αυτά σαν μια παρηγοριά βρισκόμαστε στο διαδίκτυο. Μεταδίδεται η συνεδρία στο διαδίκτυο. Colleagues. Συνάδελφοι. Contain your excitement. Αυτό συγκρατηθείτε λιγάκι αγαπητοί συνάδελφοι. Χθες έγινε συνάντηση των συντονιστών. Υπήρξε καθορισμός εισηγητών για δύο εκθέσεις, δύο εκθέσεις που πήγαν και δύο στο ΕΛΚ. Καταρχήν κανονισμός που τροποποιεί τον 261 σε σχέση με τις αποζημιώσεις προς τους επιβάτες σε περίπτωση που δεν ε, τους επιτρα... επιτράπηκε η επιβίβαση ή υπήρξε μακρά καθυστέρηση και δεύτερον πρόταση οδηγίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για την θαλάσσια χωροταξία και την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών και οι δύο αυτές εκθέσεις από το ΕΛΚ. Γνωμοδοτήσεις. Πρόταση για οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 92 του 2011 για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών σχεδίων επί του περιβάλλοντος. <clears throat> Καταρχήν δεν μας είχαν ζητήσει γνωμοδότηση, αλλά ζητήθηκε από τους συντονιστές να αποστείλουμε μια επιστολή στον Πρόεδρο και να ζητήσουμε την άδεια να εκπονήσουμε μια ε, γνωμοδότηση και θα πάει αυτή βάσει του συστήματος περιτροπής στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Για τα λοιπά θέματα οι συντονιστές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω δράση. Ανακοίνωση της Κομισιόν για την, το δεύτερο βαθμολόγιο απλοποίησης. Πρόταση για μια οδηγία σε σχέση με μέτρα για να εξασφαλιστεί υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόταση για κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό 9-12 του 2010 για, την, ε, για τον φορέα GSSS. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια <clears throat> της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ευρώπη σε σχέση με την ε, τεχνική πρόοδο για ορισμένου κανονισμούς έγγραφο εργασίας της Κομισιόν για την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες επιδοτήσεις, δημόσιες προμήθειες και κοινοφελείς υπηρεσίες. Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί ζητήθηκε από τους συντονιστές να δώσουν τα σχόλιά τους στο σχέδιο επιστολής που έχω θα αποστείλω στον κύριο Μουρέιρα της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου μέχρι την Τετάρτη 20 Μαρτίου. Για το πακέτο σιδηροδρόμου. Οι συντονιστέ έχουν εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα. και έχει καταγραφεί εκεί η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα. 7 Μαΐου είναι η δημόσια κρόαση, 8 και 9 Ιουλίου παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, 16 Σεπτεμβρίου καταληκτική προθεσμία για τροπολογίες 14 Οκτωβρίου εξέταση των τροπολογιών 26 Νοεμβρίου 26 Νοεμβρίου ψηφοφορία και έγκριση <clears throat> του σχεδίου έκθεσης στην ε, Επιτροπή μας και Ιανουάριος 2014 αν θέλει ο Θεός πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια για την ακρόαση η ακρόαση. Θα έχει δύο πάνελ, το ένα για το άνοιγμα της αγοράς και το άλλο για το πιο τεχνικά θέματα και οι συγητές του ζητήθηκε να δώσουν ονόματα δύο εμπειρογνωμόνων μέχρι την 5η 28 Μαρτίου για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε το πρόγραμμα για αυτή την ακρόαση. Για τις μελέτες για το 2013, οι συντονιστές τους έχει ζητηθεί μάλλον να προτείνουν θέματα για περαιτέρω μελέτες μέχρι το 28 Μαρτίου. Ενημέρωση του Eurocontrol για τους ενιαίους ουρανούς 2 αποφασίστηκε να προσκληθεί ο εκτελεστικός διευθυντής της Eurocontrol σε μια μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής μας, μάλλον μετά την ε, δημοσίευση των προτάσεων ΣΕΖΑ 2. Οι συντονιστές κατέγραψαν <clears throat> τα θέματα επιτροπολογιών επίσης και για τα άλλα θέματα. Ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο απήντησε στην επιστολή του κυρίου Σούλτς και ζητήθηκε από τον κύριο Σούλτς να απαντήσει τονίζοντας την ε, ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει η Κομισιόν το δικαίωμα πρωτοβουλία, εκτό αν θέλει να το εκχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον κανονισμό για τι κρατικέ επιδοτήσει. Ο κανονισμό 137 του 2007 Βάσει αυτού αποφασίσαμε να επιστήσουμε, να επιστήσουμε την προσοχή του Πρόεδρου Σούλτς στην ανάγκη να τροποποιηθεί αυτό το κείμενο με ένα κανονισμό του Συμβουλίου. Και για το φόρο στους γαλλικούς σιδηροδρόμους θα στείλω μια επιστολή στον κύριο Κάλλας και θα του ζητήσω πιο ουσιαστικές απαντήσεις και πληροφορίες. Στις 11 Απριλίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής, η συνεδρίαση της Επιτροπής μας έχει ακυρωθεί. Θυμηθείτε λοιπόν ότι στις 11 Απριλίου δεν θα συνεδριάσουμε. Αυτά λοιπόν από τους συντενιστές. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, εάν όχι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γίνονται δεκτές αυτές οι αποφάσεις των συντονιστών. Ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία για τις υπηρεσίες εδάφους. να σας πω ότι πριν ξεκινήσουμε ότι λόγω της ε, διάδοσης στο διαδίκτυο δεν υπάρχει οθόνη που να δείχνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Έχετε στο γραφείο σας, στα έδρανά σας τα αποτελέσματα και επειδή δεν υπάρχει γενική οθόνη θα αναγυγνώσκω τα αποτελέσματα και μην μου λέτε γιατί δεν επιταχύνουμε με το να παραλείπουμε τα αποτελέσματα, πρέπει να τα διαβάζω για να μπορούν αυτοί που παρακολουθούν στο διαδίκτυο να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Πάμε, <clears throat> είμαστε έτοιμοι. <clears throat> για να δούμε καταρχήν πόσοι είναι παρόντες. Κάνουμε μία ψηφοφορία ελέγχου. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλεγχος είναι αυτό, ναι. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα παραπάνω. Όχι. Πέρας. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Well, re... no, no card, no vote, I'm afraid. Όποιος δεν έχει κάρτα δεν ψηφίζει. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα παραπάνω που ψηφίζει. Okay, so Mr. Fleckenstein's highly delighted. Ο κύριος Φλακενστάν χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε λοιπόν. Πάμε συνάδελφοι. Τροπολογίες 53, 54, 55 αλλά και 57 είναι οι τροπολογίες για την απόρριψη της πρότασης Άρχεται η ψηφοφορία επί αυτών. Ηλεκτρονικά. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει ένα που παραπάνω που ψηφίζει τώρα. Και οι σοσιαλιστές έχουν πάλι ένα που ψηφίζει παραπάνω. Can an S&D substitute please remove a... Ένα αναπληρωματικός παρακαλώ να βγάλει την κάρτα του. Λοιπόν, πέρασε ψηφοφορίε, τώρα είναι εντάξει. 45 ψήφισαν, 21 υπέρ, 23 κατά. Μία αποχή, επομένως απορρίπτεται η πρόταση απόρριψης. Πάμε στο άρθρο 2, συμβαστική C. Ψήφι υπέρ. κατά αποχέ εγκρίνεται. Εκατόν εικοσιοχτώ. Ήγγιν Στεβεράκ. Και η ΙΜΚΟ 7 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 1.28 και ημικοεπτά. 7. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Είμαστε στο σωστό αριθμό. Εντάξει, κλείνει η ψηφοφορία. 27 εναντί 17 με μία αποχή γίνεται, γίνονται δεκτές αυτές τις τροπολογίες. 126 light trade. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος. Για την 126 άρχεται. Καλού κακού. Ψηφίσατε όλοι. Είμαστε μέσα στα όρια του αριθμού των βουλευτών. Πέρας. 21-19. Σας το είπα, σας το είπα. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 125 άρχεται η ψηφοφορία εδώ δεν μπορεί να δει κανεί τι γίνεται γιατί είναι όλα κυκλικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24-19 με μία αποχή γίνεται δεκτή 125. 129 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέξουμε και πάλι. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, ναι. Πέρας. 17 με 20 και μία αποχή απορρίπτεται. 130 Μπαχ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Να ελέγξουμε, βεβαίω. <clears throat> Άρχεται η ψηφοφορία για την 132. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. Πάμε στην 131 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ναι, θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι όλες πρέπει να τις κάνουμε ηλεκτρονικά πια, λέει ο πρόεδρος. Όλες. Όχι. Μα κάθε φορά όταν είναι σαφές το αποτέλεσμα λέτε να ελέγξω. 131 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Και οι αιτήσει για έλεγχο γίνονται σε εθνική βάση και όχι σε κομματική βάση. Το ΕΛΚ έχει ένα που περισσεύει πάλι. Εντάξει. Πέρασε. Απορρίπτεται. 19 με 25. 133 και 135 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 138 και 74 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτονται 1.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1.36 και 1.43 υπέρ κατά έλεγχος 1.36 και 1.43 μαζί άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 20 με 23 απορρίπτονται 1.41 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 1.39 και 1.40 μαζί. Υπέρ. Κατά. Ελεγχός. 1.39 και 1.40. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 2023 απορρίπτεται. 1.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α2 ηλεκτρονικά κατευθείαν. Α2 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, όλες. Πέρας. Δεν γίνεται δεκτή. 20-24 με μία αποχή απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α1, A1. Ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. πέρας εγκρίνεται 34 με 9 Πάμε στη σελίδα 6 στο δικό μου κείμενο και ψηφίσουμε την ΙΜΚΟ 10 για το άρθρο 1, παράγραφος 1. Σελίδα 6 στο αγγλικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Έλεγχος για την ΙΜΚΟ 10. Άρχεται. Ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-25. <clears throat> Απορρίπτει 17 του εισηγητή. Υπέρ. κατά αποχές να ελέγξουμε γιατί 17 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 22-22 ισοψηφία απορρίπτεται 195 Γκάλερ Φερμπά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε έλεγχο. Μα είναι φανερό. 195 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 15 με 28 κατά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να δει κανείς, οπότε σας κατανοώ, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να δει κανείς κυκλικά τι γίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 194. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι πέρας. 27-17 γίνεται δεκτή. 18, 18 υπέρ κατά. Άποχες εγκρίνεται. 197 εκπίπτει. Πάμε στην 10. 19 είναι η επόμενη του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 198. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 199. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.20 2.20 άρθρο 10 παράγραφος 1 υπέρ στις 220 κατά Αποχές απορρίπτεται. 2.21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 18 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος επειδή αρχίζει να κουράζεται το χέρι των ψηφοφόρων. Ήμκο 18, αυτή την ψηφοφορία. Πέρας. 43-0. Εγκρίνεται. Πρέπει να σηκώνετε το χέρι σας, το καταλάβατε αυτό. 2-23 ναι? και ήμκο 19 μαζί, ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.26 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πάμε στην 2.36. Γιατί άλλες δεν ψηφίζονται λόγω του άρθρου 50 του κανονισμού μας. 2.36. Για τα νησιωτικά αεροδρόμια. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.51 και 2.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.54 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για τη 254 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 18-26, μία αποχή, απορρίπτεται. Ήμκο 24, υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την Ήμκο 24. Άρχεται. ψηφισσατε ολοι όλοι. Πέρασε. 20-24 απορρίπτεται 2-52 υπέρ κατά Αποχέστα. θα ελέγξουμε τη 2-52 άρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε πέρας Πέρασε. 19-24 απορρίπτεται. 2-56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2-57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κεφάλαιο 4 τώρα. Συμβαστική D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ι, e, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.90. 2.95. Άρθρο 21, 295. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 297. Ήμκο 27 και 298 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 2,99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 300 υπέρ. Δεν εγκρίθηκε η 2,99, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την 300. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε για την 300. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 24 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. 302. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 304. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 304. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 30 υπέρ, 14 κατά. 305 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 305. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 26 κατά. 306 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Όντω. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 26 κατά. 307 και 308 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται 17 υπέρ 26 κατά. 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 311. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 25 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. 313 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. 18 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. 314 και ΙΜΚΟ 28 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 312 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την 316. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ, 25 κατά. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα το ελέγξω. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της Πράγματι εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ και 14 κατά. 317 τώρα. 317 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 320 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 322 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 325 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται 18 υπέρ, 25 κατά. 326 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 326 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται 38 υπέρ 6 κατά. 327 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 330 τώρα. Όχι, 329 διορθώνει ο πρόεδρος. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 330. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 331. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 332. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 333. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 333. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, 17 κατά. 37 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. όσοι θέλουν να ψηφίσουν βέβαια. Θα ελέγξουμε λοιπόν για την 37 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορίας. 36 υπέρ, 8 κατά. Εγκρίνεται. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να σηκώνετε τα χέρια σας ψηλά για να σας βλέπω όταν ψηφίζουμε. 335 και 336 τώρα που είναι οι ίδιες, μαζί ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ήμκο 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 338. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για 338 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 20 ψήφοι υπέρ και 23 κατά. 339 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 337, 340 και ΙΜΚΟ 31 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 341 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 342 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 343 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 345 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 344 και ΙΜΚΟ 32 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, τάφ, F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 422 τροπολογία τώρα, στο άρθρο 30α. Το βρήκατε? Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 425 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, ελέγξουμε για την 423 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται πράγματι. 427. Η 424 καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε 423. Αλλά υπάρχει και ΙΜΚΟ 36 που την ψηφίζουμε ως προσθήκη. Ωραία, υπέρ παρακαλώ τη ΙΜΚΟ 36. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 427 και 434. Όχι, χωριστά θα τις ψηφίσουμε γιατί πρόκειται για διαφορετική διατύπωση. 427 πρώτα λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε για την 427 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. πέρα τη φοφορία. Εγκρίθηκε 23 υπέρ 21 ψήφι κατά. 434 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για 434. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 21 ψήφοι υπέρ, 23 κατά. 426 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 430 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 431 και 432 είναι ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 433 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική G. Ζ. συμβιβαστική G. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 469 στο άρθρο 33 τώρα. Έχουμε την 469, 470, 471 και 472 που τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνονται με 29 ψήφους υπέρ και 15 κατά. Συμβαστική L τώρα. Στο άρθρο 35 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την συμβαστική αυτή τροπολογία L ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται 18 υπέρ 24 κατά, που σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες μία-μία. 493 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 495 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για 495. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 18 υπέρ 25 κατά. 494 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε για την 494. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 23 υπέρ, 20 κατά. 496, 497, 498 μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 499 καταπίπτει, 500 τώρα. 501, 502, 503, 504 ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Να ελέγξουμε άμα θέλετε, αλλά ήταν σαφές για μένα. Εντάξει, συνεχίζουμε. 505 τώρα υπέρ. 505 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 506 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 507. 508 δεν τις ψηφίζουμε. 516 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Δεν ψηφίζουν πολύ στην αίθουσα, γι' αυτό. Λοιπόν, ψηφίστε παρακαλώ τώρα ηλεκτρονικά για την 516. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 22-22 είναι το αποτέλεσμα. 509 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 509. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 18 υπέρ, 25 κατά. 510 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 511 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 512 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την 512. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 25 υπέρ, 19 κατά. 513 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 514 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 515 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την 515. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται με 22-22 ψηφία. 500 18 και 519. Έχουμε και μια προφορική τροπολογία που την βλέπετε στο κατάλογο ψηφοφοριών. Έχει κανείς αντίρρηση να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, τότε ψηφίσουμε αυτές τις δύο τροπολογίες μαζί με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 520. Αποσύρθηκε. 521 της κυρίας Βίλ. Σίπερ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 521 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε 18 ψηφίπερ υπέρ, 25 κατά. 522 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 523 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 524 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόλησης 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 30 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά. 526 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 527 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 30... Συγγνώμη. Έχουμε εδώ να κάνουμε με τον κανόνα 50. Πάμε στην απασχόληση 35. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Απασχόληση 35. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 19 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. 529 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και για την 529 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 21 ψήφοι υπέρ, 22 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. Απασχόληση 36. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε και αυτήν την τροπολογία απασχόλησης 36. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 22 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Συμβιβασ... Α, 534 πρώτα, πριν τη συμβαστική. 534 της κυρίας Τικάου, υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε 534. Ψηφίσατε όλοι. στις της 534. Απορρίπτεται 21 ψήφι υπέρ, 22 κατά. Συμβιβαστική ΆΗ τώρα γιώτα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «541 τώρα. Υπέρ παρακαλώ». Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 542. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 542. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 16 υπέρ, 25 κατά. 543 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 544 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ετυλογικές σκέψεις. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε 18 υπέρ 24 κατά. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 60. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ψηφίστε ηλεκτρονικά να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται πράγματι. 61 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και για την 61. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε 19 υπέρ 22 κατά. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 70. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορίας. Εγκρίθηκε 25 υπέρ, 17 κατά. 64 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε την 64. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Αποτέλεσμα 21 υπέρ, 21 κατά. 65 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 65. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρα της φοφορίας. 14 υπέρ, 28 κατά. Απορρίφθηκε. 66 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε για την 68 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της 18 υπέρ, 24 κατά απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για την 72 ε, ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται πράγματι 15 υπέρ, 27 κατά. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. 19 υπέρ, 23 κατά. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 77. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίες. Απορρίφθηκε 17 υπέρ 25 κατά. 2 υπέρ κατά. Ξανά. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την τροπολογία 2 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε 28 υπέρ, 13 κατά. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Συμβαστική και κάπα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε για την τριά Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 27 υπέρ 15 κατά. 81 και 82 μαζί τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε, νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 81 και 82. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκαν 25 υπέρ, 17 κατά. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απασχόλησης 2 υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την απασχόληση 2. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 17 υπέρ, 24 κατά. 84 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 87. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε 27 υπέρ, 14 κατά. 86 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά επειδή πολλοί από σας δεν ψηφίσαν, δεν σηκώσαν το χέρι, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 30 υπέρ 11 κατά. Απασχόληση 3 είναι η επόμενη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την απασχόληση. Τρία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε 18 υπέρ 24 κατά. Απασχόληση 4 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια ε, πλειοψηφία απορρίφθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 89 καταπίπτει. 90 ως προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την 90, ε, για την 90 ε, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 26 υπέρ 17 κατά. 91 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93. Ακόμα ισχύει. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 96. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις προφορίες. Απορρίφθηκε. 17 υπέρ, 23 κατά. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. απασχόλησης 6 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Απασχόλησης 6. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορία. Απορρίφθηκε. 19 υπέρ, 24 κατά. 100 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 99. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 20 υπέρ, 23 κατά. Ίμκο. 4 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά γιατί το ΕΛΚ δεν βλέπω πώς ψηφίζει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε 31 ψήφι υπέρ 10 κατά. 102 και ΙΜΚΟ 5 μαζί υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης 8 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. Την απασχόληση 8. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε 17 υπέρ 25 κατά. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και 26 6 ήταν μαζί. 104 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απασχόλησης αριθμός 1, υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την απασχόληση 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 19 υπέρ 24 κατά. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ε, νομοθετικού περιεχομένου, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, τροποποιημένη βέβαια. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 ψηφί υπέρ, 15 κατά και 10 αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ε, ψηφοφορίες. Αποτέλεσμα 19 υπέρ, 17 κατά, 8 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ζαζάρη. I Συναδελφοί, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι βέβαια διχασμένο κάπως το σώμα, αλλά αυτή είναι η απόφαση. Τώρα, συνεχίζουμε. Όσοι θέλουν να καταλήψουν την αίθουσα, ησύχω παρακαλώ, για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Κάποιος από τη γραμματεία παρακαλώ. Μπορεί να μας πει τι χάσαμε γιατί δεν ήρθανε τα καροτσάκια με το τσάι. Το επόμενό μας θέμα λοιπόν είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρημουλκουμένων τους. People, please leave. If they're not intending to stay. Όσοι παρακαλώ δεν σκοπεύουν να μείνουν για την επόμενη συζήτηση, αν έχουν την καλοσύνη να βγουν από την αίθουσα.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 Όσον αφορά την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μας κατέθεσε μία πρόταση και εγώ είμαι αρμόδιος ε, για τον τεχνικό έλεγχο των ε, μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρημουλκούμενών τους ε, και ο στόχος μας είναι βεβαίως να περιορίσουμε ή δυνατόν τον αριθμό των νεκρών από τροχαία ατυχήματα στους δρόμους και γενικότερα των ε, αριθμό των ε, τροχαίων ατυχημάτων. Ιδιαίτερα στις ε, χώρες που είναι σημεία και χώροι διαμετακόμισης, για τις χώρες αυτές είναι σημαντικό να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές, εναρμονισμένες ελάχιστες προδιαγραφές και αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνει η τεχνική ουδετερότητα, όπως την αποκαλούμε. Πάω στις τροπολογίες μου. Άρθρο 1. Σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει η δυνατότητα ε, είναι ε, όχι δυνατόν, αλλά υποχρεωτικό να υπάρχουν τεχνικές ελάχιστες προδιαγραφές για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Και πέρα από αυτό, εάν ένα κράτος μέλος ε, πιστεύει και όχι μόνο πιστεύει, αλλά πρέπει να αναγνωρίσει το ότι, όπως είπαν οι Κομισιόν και το Συμβούλιο, να υπάρξει ένας κανονισμός. Η Κομισιόν τάσεται υπέρ της ε, θέσπισης κανονισμού. Το Συμβούλιο επιθυμεί περισσότερο να θεσπιστεί οδηγία. Μία οδηγία λοιπόν η οποία θα ε, λαμβάνει υπόψη της ε, τις ε, νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν ε, στα κράτη-μέλη. Εμείς νομίζω ως Επιτροπή πρέπει να θεσπίσουμε μια ξεκάθαρη γραμμή, να πούμε ότι θέλουμε κανονισμό που να εφαρμόζεται. Και βεβαίως οι μεμονωμένες ε, αρμοδιότητες μπορούν να παραμείνουν στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά στο άρθρο 2, εκεί γίνεται λόγος για την προσαρμογή της ε, ε, ορολογίας ε, στην κείμενη νομοθεσία. 16 και 17 οι τροπολογίες μου αφορούν τον ορισμό των ενιών. Εκεί λοιπόν τίθεται κυρίως ε, το θέμα των ιστορικών οχημάτων, κατά πόσον αυτά θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ε, τεχνικούς ε, ελέγχους ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν δικές ρυθμίσεις για τα οχήματα αυτά, μόνο που θέλω να πω ότι ένα όχημα το οποίο είναι άνω των 30 ετών, το να χαρακτηρίζεται αυτό αυτομάτως ως τεχνικό όχημα δεν είναι σωστό, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία και να είναι επίσης σαφές ότι στο αμάξωμα τουλάχιστον είναι εμφανής και παραμένει εμφανής ιστορία του αυτοκινήτου. Όσον αφορά τώρα τους ελέγχους, ε, ε, πράγματι εμφανίστηκαν κάποιες ε, διαφορετικές απόψεις το δικό μου το σχέδιο μεταφράστηκε και διανεμήθηκε στους συναδέλφους. Αρκετοί εξ αυτών μου απάντησαν. Εγώ είχα ως στόχο να βελτιώσω τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αφήσω και ένα περιθώριο για ερμηνείες. Αναφέρομαι τώρα στα εξαρτήματα ενός οχήματος τα οποία έχουν τοποθετηθεί ευθύ εξ αρχής από την ημέρα κατασκευής του οχήματος αυτού. Αυτά πρέπει να παραμένουν μέχρι τέλους και το ίδιο ισχύει και για τον ειδικό εξοπλισμό, τα ιδιαίτερα ε, αξεσουάρ ενός ε, αυτοκινήτου. Τώρα, όσον αφορά στο άρθρο 4, τροπολογία υπαριθμών 19, αρμοδιότητες. Εκεί λοιπόν γίνεται περισσότερο λόγο για τα δεδομένα στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι κατασκευαστές σχετικά με τους ε, κατασκευαστές ε, των ε, εξαρτημάτων ελέγχου. Ειδική λοιπόν αναφορά στους κατασκευαστές εξαρτημάτων ελέγχου να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης ε, στα τεχνικά δεδομένα. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε ηλεκτρονική εποχή. Έτσι κι αλλιώ ε, τα αυτοκίνητα κυρίω ηλεκτρονικά ελέγχονται, γι' αυτό και αυτό που λέω είναι απαραίτητο. Τροπολογία 2021 για το άρθρο 5. Εκεί αναφέρεται η ημερομηνία ελέγχου και η πυκνότητα των ελέγχων. Εγώ λοιπόν προτείνω ε, καταρχήν να συμφωνήσουμε σε ένα ελάχιστο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι και το συμπέρασμα που προέκυψε από ε, ε, τις αναφορές των κρατών μελών για την πυκνότητα των ελέγχων. Να γίνεται λοιπόν ο έλεγχος ε, τουλάχιστον τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Τέσσερα χρόνια μετά την κατασκευή του να ελέγχεται το αυτοκίνητο και μετά ανά δύο χρόνια. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα δίκυκλα Εκεί δεν προβλέπεται βασικός ε, έλεγχος. Ε, εγώ όμως ε, στη δική μου την πρόταση, την οποία σας έχω καταθέσει, καταλήγω στις τροπολογίες 20 και 21 στο ότι τα δίκυκλα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουμε στους τεχνικούς ελέγχους. Και εδώ πρόκειται κυρίως για τις βαριές μηχανές οι οποίες ε, έχουν πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Όσον αφορά τώρα τα ρημουλκούμενα οχήματα και αυτά πρέπει να ελέγχονται εφόσον έχουν τεχνικό εξοπλισμό και ε, ζυγίζουν πάνω από 750 κιλά. Ε, την συχνότητα αυτή θα πρέπει να την καθορίσουν τα κράτη-μέλη. Τροπολογία υπερθμών 23 για το άρθρο 5. Κριτήριο mileage 160.000 χιλιόμετρα και ε, έλεγχος πριν από τα τέσσερα χρόνια. Το να συμπεριληφθούν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να το συζητήσουμε. Να δούμε μήπως ε, υπάρχει και η δυνατότητα ε, να πειραχτεί, όπως λέμε στα ελληνικά, ο δείκτης των χιλιόμετρων. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 24. Εκεί διαγράφεται ε, ο έλεγχος, μάλλον εκεί προβλέπεται έλεγχος όταν το όχημα αλλάζει ιδιοκτήτη. Για μας ε, είναι σημαντικό ο έλεγχος ε, να γίνεται στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί μετά από πέντε χρόνια. Αλλά όσον αφορά την πώληση του οχήματος καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κριτήριο ε, βελτίωσης της αξίας ε, του οχήματος και αυτό και μόνο ως κριτήριο, η βελτίωση της αξίας, ε, δεν οδηγεί στο ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος τη στιγμή που ενδεχομένω το αυτοκίνητο να είναι ηλικίας μόνο 6 μηνών. Μετά πάω στο άρθρο 12, παράγραφος ή αν θέλετε τροπολογία υπαριθμών 27. Πρόκειται για τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ελεγκτές ε, ως ε, ελάχιστο προσόν να έχουν τουλάχιστον την εκπαίδευση σε ε, εξειδικευμένο τεχνίτη και για τους μηχανικούς να προβλέπεται πτυχίο ανώτατης σχολής. Γνωρίζω ότι στα κράτη-μέλη προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες, ε, ε, στα συνεργεία ε, οι έλεγχοι γίνονται από τους συνεργάτες των συνεργείων, αλλά ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτόν που θέτει σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο και σε αυτόν που στο τέλος ελέγχει το αυτοκίνητο ως προς τη συμπεριφορά του με κριτήριο την οδική ασφάλεια, ο οποίος είναι σημαντικός για να εξετάσει ε, το σασί, τους τροχούς, ε, τον, ε, τα φρένα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, αλλά το ελάχιστο, ελάχιστο είναι να ελέγχεται το αυτοκίνητο τουλάχιστον από δύο ανθρώπους. Δηλαδή όχι αυτός που έχει κατασκευάσει το αυτοκίνητο να αποκτά ξαφνικά άλλη ιδιότητα και να γίνεται και ελεγκτής. Πάμε στην επόμενη τροπολογίας της κατεξουσιοδότησης πράξης, νομίζω ότι εκεί ε, πρέπει να προβλέψουμε την δυνατότητα εκχώρησης αρμοδίτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μόνο για πέντε χρόνια στην, ε, όσον αφορά την ε, λογοδοσία, αλλά κάθε πέντε χρόνια η Κομισιόν να αναφέρεται στους ε, περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους. Και θα μου επιτρέψετε και μια άλλη παρατήρηση, κάτι που το συζητήσαμε ως ΕΛΚ, είναι προφανώς απαραίτητο να υπάρχει ένας φάκελος για κάθε όχημα όπου αναφέρονται όλα τα σημαντικά γεγονότα που, ε, και στοιχεία που αφορούν στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει ε, και άλλα στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί κανείς να αξιολογήσει καλύτερα το αυτοκίνητο και να μην υπάρχει δυνατότητα να πειραχτεί όπως σας είπα ε, ο συνολικός αριθμός των χιλιόμετρων. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν μαζί μου για όλα αυτά τα θέματα. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να κατατεθούν τροπολογίες, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και εγώ λοιπόν προφανώς ε, έλαβα υπόψη μου την πρόταση Κομισιόν και κατέθεσα τις δικές μου τροπολογίες. Προσβλέπω στην εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όπως είπε ο κύριος Κούνο, συνεισηγητής. Το πακέτο αυτό για την αξιοπιστία των οχημάτων είναι ακόμα ένα κεφάλαιο που αφορά τους στόχους για την οδική ασφάλεια μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. και το όραμά μας για το 2050 σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων του περιβάλλοντος. Εγώ είμαι υπεύθυνη για το τμήμα των επιθεωρήσεων των οχημάτων για τα θέματα αυτά και για μένα το θέμα αυτό των ελέγχων και επιθεωρήσεων των οχημάτων θα πρέπει να συνάδει με την καλύτερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των επιθεωρητών και την επιβολή σαφών κανόνων από τα κράτη-μέλη. Θέλω εδώ να κάνω μια σύντομη εισαγωγή στις τροπολογίες μου για αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει σαφές <clears throat> τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί οχημάτων γίνονται και για άλλους ε, κοπούς. Παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για ταχογράφους. Ο κύριος Κούν ανέφερε την ε, έννοια των τεχνικών ελέγχων και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί η πρόταση της Κομισιόν για μένα θεωρείται, για μένα είναι απόλυτα επαρκής. Τι ακριβώς σημαίνει επίσης επιχείρηση μεταφορών στον τομέα αυτό, ο οποίος θα αντιμετωπιστεί από αυτή την ε, έκθεση. Τονίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή αυτών των ελέγχων στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό των οχημάτων τα οποία δεν <clears throat> συμμορφώνονται με τις ε, υποχρεώσεις αυτές ξεκινάνε από 0,3% και φτάνουν 63% σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτές οι διαφορές μπορούν να είναι τεράστιες και μεταξύ γειτονικών χωρών. Μερικές χώρες έχουν πάρα πολύ ενδελεχείς διαδικασίες ε, ελέγχων που είναι παρόμοιε αυτών των περιοδικών ελέγχων οχημάτων. Άλλες χώρες ελέγχουν ελάχιστα ή μόνο την, ε, τα έγγραφα του οχήματο. Γι' αυτό για μένα η επιλογή των οχημάτων που πρέπει να υπόκειται σε αυτού του τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται στο προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων μεταφοράς. Πρέπει εμείς να ανταμείβουμε αυτούς οι οποίοι διατηρούν σε καλή κατάσταση τον στόλο οχημάτων τους με τακτικούς ελέγχους. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Πιστεύω θα ήταν θετικό να εφαρμοστεί σε δύο στάδια και γι' αυτό προτείνω για το άρθρο 24 να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό μέσα σε τρία χρόνια για τα οχήματα πάνω από 3,5 τόνους και πέντε χρόνια για αυτά που είναι κάτω από 3,5 τόνου, Από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό ο κανονισμός. Επίσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τεχνικοί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται χωρί καμία διάκριση επί τη βάση της εθνικότητα του οδηγού ή του αριθμού της ε, πινακίδας του αυτοκινητού. Προτείνω λοιπόν μια σειρά από τροπολογίε για το άρθρο 8 και εδώ τονίζω ότι πρέπει η κατάρτιση να είναι το βασικό στοιχείο αυτού του συστήματο και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απώλειες χρόνου για τις επιχειρήσεις και ε, ατέλειες στο σύστημα. Και για το εύρος εφαρμογής θεωρώ ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα κάτω από 3,5 ε, τόνους, όπως και τα παρελκόμενά τους τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για εμπορικούς στόχους στις οδικές μεταφορές και δεν βλέπουμε να μειώνονται τα ατυχήματα, τα ποσοστά ατυχημάτων για αυτά τα οχήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή αυτών των ελέγχων επίσης και για τα τρακτέρ κατηγορία TAF 5, διότι αυτά τα οχήματα πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθούν οι προδιαγραφές για βαρέα εμπορικά οχήματα. Υποστηρίζω πλήρως την ε, ενοποίηση των ε, κανόνων για την ε, σωστή φόρτιση των οχημάτων και την σωστή ασφάλιση του φορτίου, γιατί αυτό οδηγεί σε 25% των ατυχημάτων και επίσης πρέπει να υπάρχει έλεγχος για υπερβολική φόρτωση αυτών των οχημάτων. Πρέπει επίσης να διαλευκανθούν οι ευθύνε για την τεχνική κατάσταση των οχημάτων. Γι' αυτό προτείνω τροπολογίε στο άρθρο 7, όπου πρέπει να γίνει σαφέ ότι οι μεταφορεί που χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα θα πρέπει να είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφαλεία. Και το ίδιο αφορά για την ασφάλιση του φορτίου στα οχήματα. Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, <clears throat> αλλά πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για περίπτωση ατυχήματος στους ελέγχους αυτούς που γίνονται στο δρόμο για τα οχήματα μαζεύουμε πολλά δεδομένα τα οποία νομίζω ότι μετά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει ένα σύστημα καθορισμού κινδύνου για το μέλλον. Τώρα σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία και περιμένω να ακούσω και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ, Λεωπρόεδρος. αγαπητοί συνάδελφοι. Ήμουνα και εγώ εισηγήτρια για το τρίτο τμήμα του πακέτου αυτού, που βέβαια ήταν το πιο μικρό, όχι όμως και το λιγότερο σημαντικό. Πρόκειται για την καταχώρηση και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να συνοδεύουν ένα όχημα. Στόχος της καταχώρησης είναι κάθε όχημα να διαθέτει κάποιο πιστοποιητικό το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια που κυκλοφορεί στους δρόμους μας. Η διαδικασία βέβαια καταχώρησης των οχημάτων πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζει ε, οχήματα που να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφάλειας. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάνω απ' όλα είναι στα διάφορα πιστοποιητικά που συνοδεύουν την καταχώρηση να αναφέρονται όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί προσωρινά ή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να καταργηθεί μια τέτοια καταχώρηση. Εφόσον δηλαδή γίνει κάτι που καταργηθεί αυτή η καταχώρηση, τότε δεν θα πρέπει να επιτρέπεται και η κυκλοφορία του οχήματο στους δρόμους μας. Πάντως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι την μεταφορά ε, σε καταλόγους καταχώρησης άλλες χώρες, εφόσον το όχημα μετακινηθεί και κυκλοφορεί μόνιμα πια σε μια άλλη χώρα. Και αν βρεθούν ε, αδυναμίες ή ε, απάτες θα πρέπει να αποσυρθεί το πιστοποιητικό και να μην επιτρέπεται πια η καταχώρηση του οχήματος αυτού. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά Στηρίζω πρέπει να ξέρετε την πρόταση, πάντως προτείνω συγχρόνως και κάποιες τροποποίησεις προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άχθος και να γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή της πρότασης αυτής. Να μειωθεί για παράδειγμα ε, ο όγκος των ε, πιστοποιητικών που χρειάζονται, των εγγράφων που πρέπει να φέρουν ή οδηγοί για να γίνεται η καταχώρηση αυτή. Επίσης, Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2005, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου του οχήματος. Επιπλέον, ο, ο ηλεκτρονικός κατάλογος καταχώρησης είναι κάτι που βρίσκουμε απόλυτα λογικό και θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος να συνδεθούν όλες οι βάσεις δεδομένων των διαφόρων χωρών μελών σε όλες τις χώρες ε, μέλη πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και επαρκής καταχώρηση. Τι γίνεται όμως όταν ε, πουληθεί το όχημα. Ο ιδιοκτήτης μερικές φορές πρέπει εκείνος να φροντίσει να αφαιρεθούν τα δεδομένα από την καταχώρηση σε μια χώρα για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ε, θέλουμε μετά από πέντε χρόνια να υπάρξει αναθεώρηση. Τέλος, ευχαριστώ πολύ σε όλους τους συνεισηγητές και είμαι στη διάθεσή σας ε, βεβαίως για ό,τι τροπολογίες θα θέλατε ενδεχομένω να υποβάλλετε στην πρόταση αυτή. Ε, ευχαριστώ. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για την ε, αξιοπιστία των οχημάτων στο δρόμο. Το τα κακά νέα είναι ότι έχω άλλους 15 ομιλητές. Ο κύριος Ρανοτσάριο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Gross, Bangen και τα λοιπά. Duran. Mr. Perker, Mrs. Foster, Mr. Van Dalen, Mr. Ferber, Mrs. Griesbeck, Mrs. Tico and Mr. Back and myself. Anybody else? I don't think there's Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Νομίζω ότι όλοι που είναι εδώ θα μιλήσουν. Εντάξει. Δύο λεπτά ο καθένας, <clears throat> αλλιώς δεν τελειώνουμε ποτέ. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ο κύριος Τσάρε, ελπίζω να το έχω πει σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Ήμουνα ο εισηγητής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το πακέτο αυτό για την ε, αξιοπιστία των οχημάτων. Κάποιες ε, ανησυχίες μας τώρα για το θέμα αυτό. Ξεκινάμε από τη νομική μορφή του νομοθετήματος. Εμείς υποστηρίζουμε τον κανονισμό αυτό που προτείνει η Κομισιόν που ως ήπια νομοθεσία αφήνει και κάποιο περιθώριο επιλογής στα κράτη-μέλη. Αν πάρει τώρα το χαρακτήρα μιας οδηγίας νομοθεσία θα καθυστερήσουμε τη διαδικασία αυτή. Και σε σχέση με την εκθεσή σας, εκτιμώ την έκθεση του κυρίου Κούν που περιλαμβάνει τα σκούτερ και τα μοτοποδήλατα στη, στη σφαίρα εφαρμογής αυτής της έκθεσης. Είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες των δρόμων φυσικά. Και συμφωνούμε με τον εισηγητή σας ότι η συχνότητα 4-2 πρέπει να 4-2-2 και όχι 4-2-1 για αυτά τα οχήματα για το γεγονός έχουν, επειδή έχουν μικρότερη, ε, μικρότερο αριθμό χιλιόμετρων που καλύπτουν κάθε χρόνο. Αλλά εμείς από την άλλη πλευρά έχουμε πολλές αμφιβολίες σε σχέση με την θέση σας που ζητάτε να ακυρωθεί η πρόταση που λέει ότι ένα αυτοκίνητο που φτάνει τα 160.000 χιλιόμετρα στο πρώτο τεστ του θα πρέπει να υπόκειται σε ελέγχους κάθε χρόνο. Θεωρούμε πρέπει να διατηρήσουμε το 4-2-2 και όχι το 4 ότι όλα τα οχήματα που καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο θα πρέπει να την χάνουν πιο συχνών ελέγχων. Γιατί σίγουρα είναι πιο μεγάλος ο κίνδυνος ατυχήματος και για να είμαι ειλικρινής υπάρχει ο κίνδυνος μεν χειραγώγησης στα όργανα του οχήματος, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην δεχτούμε αυτή την πρόταση. Και σε σχέση με την ε, σύγκρουση διαφόρων προτάσεων, εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την έκθεσή σας. Μόνο μια μικρή πρόταση για τους ελέγχους αυτούς γιατί βλέπουμε ότι η Κομισιόν μας ζητάει ένα ποσοστό 5% όλων των οχημάτων να ελέγχεται, αλλά αν σκεφτείτε το μεγάλο αριθμό των ελαφρών εμπορικών οχημάτων που κυκλοφορούν, τότε ο στόχος αυτός είναι υπερφιλόδοξος και μη εφικτός γιατί τα ελαφρά οχήματα είναι πάνω από 80% των συνολικών εμπορικών οχημάτων τα ελαφρά που κυκλοφορούν. Αναρωτιόμαστε λοιπόν κατά πόσο είναι καλή ιδέα να ζητήσουμε να υπάρχει επίσημα έλεγχος και ίσως μπορούν τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους τους για να πετύχουν τους στόχους τους. Έχουμε και ένα όραμα στην Επιτροπή μας. Να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ε, συμμόρφωσης προς τις υποδιαγραφές που να αντικαταστήσει το εθνικό ε, πιστοποιητικό. Νομίζω ότι αυτά που αναφέρεται στο άρθρο 10β στην έκθεση του κ. Κούν είναι ένα πρώτο βήμα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και γι' αυτό χαιρόμαστε για την πρότασή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο λεπτά ο καθένα, παρακαλώ. Ε. Ο κύριο Μπένιν πρώτο, ο οποίο πρέπει να φύγει να πάει να ψηφίσει αλλού και μετά γρό. Παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ. Πράγματι και εγώ είμαι ικανοποιημένο από τη γενική προσέγγιση των εισηγητών όσον αφορά για τις, τους περιοδικούς αυτούς ελέγχους. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση ενός ενιαίου χώρου μεταφορών στην Ευρώπη, που είναι ισχύει ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως αυτές οι απαιτήσει δεν θα πρέπει να επισκιάζουν τους ελέγχους σε όλα τα οχήματα, είτε γίνονται περιοδικά είτε όχι. Γι' αυτό και χρειάζεται κάποια καλή ισορροπία ανάμεσα στους εθνίδιους ελέγχους και τους περιοδικούς ελέγχους. Εγώ δεν βλέπω εδώ γιατί να βάλουμε τα μικρά και μεσαία ε, ρημούλκα. Φοβάμαι ότι μερικές φορές μπορεί να είναι λάθος να λάβουν υπόψη μας το μέγεθος των ε, ρημουλκόμενων. Έπειτα, όσον αφορά την ασφάλεια του φορτίου, εγώ δεν θα έβαζα εξαίρεση στους ε, ευνίδιους ελέγχους για την περίπτωση αυτή των φορτίων. Πρέπει να δούμε όμως πού θα γίνεται αυτός ο έλεγχος ακριβώς. Είναι πρακτικό δηλαδή το ζήτημα. Πάντως το πιο σημαντικό για μένα είναι οι τροπολογίες 5 και 28 που αναφέρονται στην διάρθρωση των ελέγχων στις χώρες μέλη. 10 χώρες έχουν τέτοιους ελέγχους. 10 από τις 27 χώρες έχουν συστήματα δηλαδή όπου τα γίνονται και στα φορτία οι έλεγχοι και τρεις ε, από τις καλύτερες περιπτώσεις έχουν ε, καλά τέτοια μοντέλα. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να συμφωνήσω με τον εισηγητή για την υποχρέωση διάκρισης των ελέγχων στα φορτία και στα οχήματα σε όλες τις χώρες μέλη. Ναι, ναι, τελειώνω. Αυτό είναι ήταν το κυριότερό μου, οπότε σταματάω εδώ. Ναι, το δικό Κοιτάξτε. χρόνο πέραν Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για, τις, ε, για την έκθεσή του. Ε, βεβαίως ε, εμείς στο ΕΛΚ μελετήσαμε την έκθεση του αδέλφου κυρίου Κούν και όπως ξέρετε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να υπάρχει υπεραξία σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Εμείς προερχόμαστε από μια συνοριακή μεθοριακή περιοχή και γι' αυτό η διασυνοριακή συνεργασία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταργήσουμε τα σύνορα, αυτό όμως σημαίνει για μένα τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, πρέπει να επιδιώξουμε υψηλέ προδιαγραφές ποιότητας, γιατί αυτή είναι η βάση της αμοιβαία αναγνώρισης. Και αυτή η οδηγία δεν μπορεί να επιτρέψει να επιδεινωθεί η ποιότητα. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν δύο κριτήρια, αφενός η ασφάλεια και φετέρου η προστασία του περιβάλλοντος. Και το τελευταίο είναι θα πρέπει να υπάρχει προοπτική να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή λαθροχειρίας. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε καλά δίκτυα ενημέρωσης. Ε, θεωρώ ότι πρέπει πέρα από το κράτος να προστατεύσουμε κυρίως τον πολίτη όχι τα δεδομένα. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι σωστή. Όσον αφορά τη δική μου τη χώρα, να σας πω μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Δηλαδή έχουμε το περίφημο διαβατήριο του αυτοκινήτου, το Car Pass. Και αυτό λοιπόν το διαβατήριο σας ενημερώνει για τη ζωή του αυτοκινήτου, τον αριθμό των χιλιόμετρων και επίση και το διαβατήριο αυτό θα μπορεί να δώσει και πληροφορίε για τα βαριά ατυχήματα στα οποία έχει εμπλακεί το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν μην ξεχνάτε ότι ε, στα αυτοκίνητα δίνονται μέχρι και 40% λανθασμένες πληροφορίες. Με αυτή λοιπόν την πρωτοβουλία επιτυγχάνουμε προστιθέμενη αξία για τον πολίτη, για την ασφάλεια, για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τα άλλα τα υπόλοιπα θέματα σε αυτά θα αναφερθούν οι συνάδελφοι. Η κυρία Ντουιρόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις πτυχές στο θέμα αυτό καταρχήν στην έκθεση του κυρίου Κούν είναι το θέμα της συχνότητας των ελέγχων. Εγώ υποστήριζω το 4-2-1, αλλα και το θέμα της απόστασης που έχει διανύσει ένα όχημα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Είναι σαν να λέμε ότι για να μην έχει κανεί πυρετό πετάμε το θερμόμετρο. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και η απόσταση που διανύει ένα αυτοκίνητο. Αν κάποιοι χρησιμοποιούν μόνο για λίγα χιλιόμετρα τα οχήματα, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να έχουμε μια διπλή λοιπόν κλίμακα, ηλικία και χιλιόμετρα που έχει διανύσει ένα όχημα. Αυτό θα ήταν καλύτερο για να έχουμε ενιαία κριτήρια. Δεύτερο θέμα, το θέμα της ανεξαρτησίας των ελέγχων στα συνεργεία. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ε, ανεξάρτητους φορείς. Αυτό ε, μπορεί να δίνει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχει σχέση αιτίου και αιτία του. Ίσως είναι άλλοι λόγοι που οδηγούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους. Εγώ νομίζω ότι η ανεξαρτησία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορεί ο γιατρός να είναι και φαρμακοποιός ε, συγχρόνως. Και τέλος, για τα θέματα του περιβάλλοντος, νομίζω ότι η έλεγχη για την εκπομπή σωματιδίων και οξυδίων του αζότου δεν είναι επαρκές να βασιζόμαστε μονάχα σε συστήματα τα οποία βρίσκονται μόνο πάνω στο όχημα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτήν την ε, τεχνολογία θα πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι ανεξάρτητοι <clears throat> ακόμα και αν για τα νέα οχήματα είναι τόσο λεπτά τα σωματίδια και οι εκπομπές που είναι πολύ δύσκολο να τα ελέγχουν. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ που μένετε μέσα στα χρονικά σας όρια. Κυρία Ροσεμπάχ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεση κυρία Κούν. Η ομάδα μου έχει διαφορετικές απόψεις γιατί υπάρχουν ε, διαφορετικά συμφέροντα αλλά από τη δική μου πλευρά εγώ συμφωνώ με τον Ματέο Γκρός και εγώ έρχομαι από μια χώρα που υπάρχει πολύ διαμεθοριακή κυκλοφορία οχημάτων για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινέ <clears throat> ρυθμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιοδήποτε όχημα, από όποια χώρα και να έρχεται, θα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες γενικής ασφάλειας του οδικού χαρακτήρα και γενικών προτύπων. Δεν μπορώ να καταλάβω να έχω αυτοκίνητα τα οποία έρχονται και τα οποία δεν έχουν καλά φρένα ή δεν λειτουργούν τα φώτα τους και όλα αυτά. Αυτό επομένως πρέπει να ισχύει για όλα τα οχήματα και αυτό ισχύει και για τα τρακτέρ τα οποία πολλές φορές καταλαμβάνουν μια μισή λωρίδα στο δρόμο και αναγκάζουν πολλά αυτοκίνητα να κάνουν επικίνδυνα πράγματα. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και ρύθμιση στα θέματα αυτά. Και τα μικρά, τα, ελαφρά ε, εμπορικά οχήματα, τα βαν, θα πρέπει και αυτά να, κατα... να ελέγχονται. Πολλές φορές έρχονται στο δρόμο και τρέχουν με 180 χωρίς να έχουν καν ασφαλίσει το φορτίο του. Λοιπόν, Επομένως, νομίζω ότι είναι λογικό να εφαρμόσουμε το 422. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα μοτοποδήλατα και τα σκούτερ, οι βέσπες, περιλαμβάνονται σε αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχουν συμφωνίες για να περιορίζεται η ταχύτητα των οχημάτων, αλλά όταν αυτό το όριο είναι μονάχα 300 300 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό δεν ωφελεί καθόλου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παντού ότι έχουμε τα ίδια στάνταρ ασφαλείας. Mr. two minutes, please. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή που έγινε και επιτρέψτε να αφαιρθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Όπως και πολλοί άλλοι, θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε τους ελέγχους και στα ε, δίκυκλα, γιατί υπάρχουν και τα σχετικά στατιστικά δεδομένα. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα αφορούν τα δικύκλα. Ένα άλλο θέμα είναι η συχνότητα των τεχνικών ελέγχων. Ποια είναι δηλαδή η δική μας άποψη. Το 4-2-2, δηλαδή 4 αρχικά τεσσερα αρχικα από την ημερομηνία κατασκευής και μετά ενα δύο χρόνια, αυτό είναι μια καλή λύση από το να πρέπει κανείς να ε, πηγαίνει σε έλεγχο κάθε χρόνο. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κοινωνική διάσταση του θέματος. Ε, και δεν πρέπει να υπάρξει απαραίτητα κοινωνική επιβάρυνση τη στιγμή που σήμερα ο τεχνικός εξοπλισμός των αυτοκινήτων επιτρέπει να γίνεται ο έλεγχος κάθε δύο χρόνια. Το επόμενο επίμαχο θέμα είναι κατά την άποψή μου η, πρόταση της Κομισιόν. Δηλαδή όταν το αυτοκίνητο θα έχει διανύσει 160.000 χιλιόμετρα από εκεί και πέρα να ελέγχεται κάθε χρόνο. Συμφωνούμε με αυτό. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι οι προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τα προσόντα των ελεγκτών. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές και να μπορεί ο έλεγχος ε, να είναι και ένα είδος τουρισμού με την έννοια δηλαδή ότι να μπορεί να πάει κανεί σε διπλανό κράτο που έχει λιγότερε προδιαγραφέ και λιγότερο αυστηρέ προδιαγραφέ για να αποκτήσει από εκεί την έγκριση τεχνικού ελέγχου. Γνωρίζω βεβαίω ότι στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Παραδείγματο χάρη, οι συνάδελφοί μα από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, στηρίζουν το ότι τελικά ε, εκείνος που επισκευάζει το αυτοκίνητο να μπορεί να κάνει και τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι ε, με τον τρόπο αυτό προφανώς και υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Ο κύριος ε, Πέρκα. Πέρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές γιατί πράγματι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας ενδιαφέρει. αυτό είναι ο στόχος μας, ε, να υπάρχουν τακτική, ε, τεχνική έλεγχη και λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα επί των οποίων δεν συμφωνούμε. Εγώ θα ήθελα να αφαιρθώ στο θέμα των τεχνικών ελέγχων. Ο κύριος Κούνες στην τροπολογία υπαριθμών 5 προτείνει ότι η επιχειρήσεις, οι κατασκευαστές να μην μπορούν να κάνουν τους τεχνικούς ελέγχους. Πιο απλά, αυτοί που κάνουν ε, την ε, συντήρηση αυτοκινήτου να μην μπορούν να κάνουν και τον έλεγχο. Να σας πω τι γίνεται στην Αυστρία. Όσον αφορά τον αριθμό των τροχιών οτυχημάτων, εμείς τα πάμε πολύ καλύτερα από άλλα κράτη-μέλη, γιατί έχουμε διαφορετικό σύστημα ελέγχου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 6% των τροχιών οτυχημάτων ανάγεται σε τεχνικής φύσεως προβλήματα. Στην Αυστρία όμως το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 2%. Ε, σε εμά υπάρχει η δυνατότητα όταν πάει κανείς το αυτοκίνητό του για συντήρηση να κάνει και τον τεχνικό έλεγχο. Όμως είναι δύο διαφορετικές μονάδες και αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους επιβάλλονται αυστηρές κοινώσεις. Και ο ελεγκτής, εάν ε, διαπιστωθεί ότι προέβη σε ολιγορία, του αφαιρείται η άδεια. Άρα δηλαδή, καταλαβαίνετε, το σύστημα είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ απευθύνομαι στον κύριο Κούν να αποσύρει ε, την τροπολογία του, δηλαδή ότι πρέπει απαρέγκλητα να υπάρχει διαχωρισμός ε, του ελέγχου, ε, να μην μπορεί ο κατασκευαστής και ε, ο ελεγκτής ε, να βρίσκονται στην ίδια μονάδα. Να το αποσύρει αυτό, γιατί ξέρετε αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δική μου την πατρίδα. Πάρα πολλές μονάδες ε, θα αναγκαστούν να κλείσουν. Δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ ή δυνατόν να αποσύρετε αυτή σας την τροπολογία. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές και όλοι συμφωνούμε βέβαια ότι θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο ασφαλείς ε, δρόμους και να έχουμε ασφαλή οχήματα όσο γίνεται πιο πολύ. Για την έκθεση Κούν. Είναι καλό που βλέπουμε ότι αναφέρονται εδώ τα παλιά οχήματα, δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Όσον αφορά τα ρημούλκα, εμεί δεν πιστεύουμε ότι τα μεσαία και τα μικρά πρέπει να συμπεριληφθούν. Όσον αφορά τα εμωτή, έχουμε ένα σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο που όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα χιλιόμετρων, είναι θέμα ηλικία. Από τα τρία χρόνια και μετά, κάθε όχημα πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο. Και αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε. Δεν ε, βλέπουμε βέβαια να υπάρχει και πρόβλημα αν άλλε χώρε έχουν ένα άλλο σύστημα που να ισχύει. Έχουμε 20.000 μικρές επιχειρήσεις και 50.000 επιθεωρητές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τη δομή. Εδώ είναι λοιπόν που έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μιλάμε για ρυθμίσεις και πώς θα πετύχουμε περισσότερη ελαστικότητα και επικουρικότητα. Αυτό πρέπει να λυθεί. Όσον αφορά τι κατεξουσιοδότηση πράξη, το ίδιο ισχύει. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση τη κυρία Αναμόβερ. Εδώ για το εύρος εφαρμογής. Όταν κοιτάμε τα περί πρέπει να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε τους ελέγχους στα μεγάλα οχήματα και αν δεν υπάρχουν ε, οι πόροι για να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί, δεν θα λειτουργήσει και το σύστημα. Συμφωνώ με τον κύριο Μπένεν τώρα για τα τρακτέρ. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να ελέγχουμε το ρόλο τα τρακτέρ. Όσον αφορά τώρα τα πιστοποιητικά. Ναι, αν πρόκειται για τον οδηγό, ναι, αλλά αν ας πούμε έχει κλαπεί το όχημα, τέλος. Τι χρήματα θα πάνε στην, ε, στον έλεγχο της ασφάλειας. Αν πρέπει να προσθεθεί αυτό στα διόδια, δεν συμφωνούμε. Τώρα για την άλλη έκθεση. Το σύστημά μα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας ικανοποιεί, δεν θέλουμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή όταν βγαίνει από το δρόμο για κάποιο χρονικό διάστημα το όχημα, δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Και για την σύνδεση ηλεκτρονικών δεδομένων πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα χωρίς να προσθέσουμε υπερβολικό κόστος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντάλιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, με εκπλήσει και εμένα. Άκουσα την συζήτηση αυτή όσον αφορά την ασφάλεια στους δρόμους. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμα υπάρχουν πολλές αποκλήσεις. Εμείς θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να λειτουργήσει τέλεια. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως γιατί να πάμε σε ένα νέο σύστημα τη στιγμή που έχουμε ένα το οποίο ήδη λειτουργεί. Οι έλεγχοι στους δρόμους, οι ευνίδοι υπάρχουν, αλλά αν θέλουμε να τους ενισχύσουμε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε παραπάνω ε, ελέγχους, παραπάνω οχήματα στους δρόμους, τις αστυνομίες που θα κάνει τους ελέγχους κλπ. Οι έλεγχοι τώρα, κατά πόσο γίνονται στα συνεργεία ή όχι. Οι έλεγχοι αυτοί μέχρι τώρα γίνονται καλά. Λειτουργεί πολύ καλά το σύστημα. Όλοι είναι ικανοποιημένοι. Οπότε, Πρόεδρε, δεν βλέπω. Φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε τεράστια φούσκα εδώ για να αλλάξουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά. Όσον ε, αφορά τώρα τις ε, μηχανές, και αυτό νομίζω ότι μέχρι τώρα λειτουργεί καλά. Και δεν βλέπω γιατί πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πολλές περίεργες ιδέες εδώ πέρα διαβάζω για τα 160.000 χιλιόμετρα για παράδειγμα. Πρόεδρε, Ε, η ίδια θα λέει η Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της. Ευχαριστώ, ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την άποψή μου ως σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Και εδώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα, είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα κανονισμό ή θα ήταν καλύτερο να γίνει μια οδηγία Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για το αν είναι καλύτερο να έχουμε ένα κανονισμό ή μια οδηγία ή αν μπορούμε πολλά από αυτά τα θέματα να τα αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Το δεύτερο έχει να κάνει με την επέκταση των κατηγοριών οχημάτων για τους ε, οδικούς ελέγχους οι στατιστικές στατιστικές δεν ε, δικαιολογούν <clears throat> το να γίνει κάτι τέτοιο να υπάρξει και το θέμα αυτό. Οι γενικοί έλεγχοι βέβαια πρέπει να ισχύουν, αλλά για τους ελαιοδικούς ελέγχους το θέμα είναι για τα ελαφρά οχήματα. Επίσης το θέμα της συχνότητας των ελέγχων. Ιδίως όταν ένα όχημα έχει κάνει ήδη ένα τεχνικό έλεγχο, ίσως θα πρέπει να γίνεται πιο απλά ο οδικός έλεγχος. Από τα θέματα βέβαια της ασφαλείας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα τηρούνται και θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο θέμα του φορτίου και της ασφάλισης του φορτίου από ότι για την ε, ποιότητα του αυτοκινήτου. Για τα οχήματα τώρα, εγώ άμα δω παραδείγματος το θέμα της Αυστρίας στην, ε, για το θέμα των οχημάτων που είναι πάρα πολλά τα φορτηγά τα οποία κυκλοφορούν σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν ε, ταξινομηθεί σε αυτή τη χώρα, όπως γίνεται στην Αυστρία ή στη Δανία σε άλλα θέματα. Σίγουρα δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε με μια τέτοια νομοθετική πράξη τα θέματα της ε, ε διαμετακόμισης. Νομίζω ότι ένα όχημα μπορεί να το... Ένα φορτηγό μπορεί να ελεγχθεί 4 ή 5 φορές. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Για τα θέματα της ταξινόμησης έχω πολλές ε, αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν με τον τρόπο αυτό θα επιτρέψουμε κάποιον να περάσει από μια χαμηλή κατηγορία σε μια καλή, καλή κατηγορία και δεν ξέρω αν αυτό θα επιτρέπει στους ελεγκτές να παρακολουθούν στο διηνεκές της εταιρείες. Κυρία Γκρίσπεχ. Κυρία Γκρίσπεχ, δύο λεπτά. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Άκουσα, σκέφτηκα μετά από όλα αυτά που άκουσα. Στο λίγο χρόνο που έχω θα σας πω το εξή. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την κυρία Ζινάνοβα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες για το ότι συμφωνώ με πολλά σημεία, όπως το θέμα της κατάρτισης, το θέμα των απαιτήσεων ε, για προσόντα, αλλά θα περιοριστώ σε κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την τροπολογία 5 στην έκθεση για τον σε βάθο έλεγχο, δηλαδή σε περίπτωση που ο αρχικό έλεγχος δεν είναι ικανοποιητικό, τότε να γίνεται πιο προθυμένος έλεγχος, είτε από κινητέ μονάδες, είτε μέσω κέντρων ελέγχων που θα βρίσκονται εκεί κοντά, λέει το κείμενο με πολλούς συναδέρφους και εγώ συμφωνώ να υπάρχει εναρμόνιση, αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι στις χώρες μας έχουμε κάποια οργάνωση όλοι για ελέγχους που λαμβάνουν υπόψη περιορισμούς γεωγραφικούς, διαθετικούς κτλ. Για παράδειγμα, από τη δικιά μου χώρα που γνωρίζω κάπως καλύτερα, στη Γαλλία έχουμε 500 εγκεκριμένα κέντρα τεχνικού ελέγχου που κάνουν και ελέγχους στα βαρέα οχήματα, αλλά πολλές φορές βρίσκονται πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να γίνονται κανονικά οι τεχνικοί έλεγχοι. Δεν έχουμε κινητές μονάδες τεχνικού ελέγχου και εδώ συμφωνώ με αυτού που μιλάνε για την επικουρικότητα και δεδομένου του κόστου μια τέτοια κινητή μονάδα τη σήμερον ημέρα μάλιστα, είμαι πολύ επιφυλακτική. Έπειτα, συμφωνώ με τον κύριο Γκρό για το ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το χαρτί που μπορούμε να παίξουμε στι διασυνοριακέ περιοχές. Εκεί δηλαδή που ε, υπάρχει σταυροδρόμι μεταξύ πολλών χωρών, πρέπει να δούμε το άρθρο 19 και την τροπολογία που προτείνεται εκεί. Τέλος, στα πλαίσια του σε βάθος ελέγχου να λάβουμε υπόψη μας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όταν, δηλαδή για τα φρένα, για τα ελαστικά και να λάβουμε υπόψη μας πάντα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστούμε κυρία Τικάου τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να στηρίξω αυτά που είπε νωρίτερα ο κύριος Έρτοκ για τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο. Νομίζω κι εγώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θέλω να αναφερθώ επίσης και στην έκθεση της κυρίας Άβυζα. Είναι σημαντικό να μειωθεί το διοικητικό άχθος και είναι σημαντικό επίσης η έλεγχοι αυτοί να αναγνωρίζονται αμοιβαίως από όλες τις χώρες μέλη. Επίσης, άπαξ και πολιθεί το όχημα και πριν καταχωρηθεί εκ νέου, πρέπει να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη για το όχημα αυτό. Γιατί έτσι όπως είπε και η συγκήτρια, η ευθύνη αυτή δεν ε, καθορίζεται σαφώς. Πάντως δεν συμφωνώ ότι είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ο οποίος μπορεί να ακυρώσει το πιστοποιητικό καταχώρησή του. Είναι επικίνδυνο γιατί αν έχει υπάρξει ατύχημα το άτομο αυτό μπορεί να κυρώσει το πιστοποιητικό του. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο. Αυτή τη δυνατότητα δεν πρέπει να την έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων. Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ χρήσιμο να μειώσουμε το διοικητικό άχθος μέσω ενός κοινού εντύπου. Θα μειωνόταν έτσι η γραφειοκρατία και θα διευκόλυνε και τους ευνίδιους ελέγχους. Τέλος, θέλω να σας πω πως στηρίζω την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Να υπάρχει σύνδεση δηλαδή μεταξύ αυτών. Και όσον αφορά την ηλεκτρονική καταχώρηση, η προθεσμία ήταν στα τέλη του 2012. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ηλεκτρονικών αυτών ε, ε, καταλόγων καταχώρησης. Κάποιες χώρες έκαναν κάποια βήματα, κάποιες άλλες όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει τις διαδικασίες επί παραβάση εναντίον των χωρών που δεν έχουν προχωρήσει. Χρειάζεται όμως να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακούγοντας αυτά που ελέγχθησαν, όλοι λένε ε, ότι έχουν τους καλύτερους όρους στη δική τους την πατρίδα. Ε, τότε γιατί συζητάμε. Εγώ όμως δεν σκέφτομαι έτσι. Και εγώ έρχομαι από μια μικρή χώρα. Ε, όπως είπε ο πρόεδρος Διακόπτας, το ίδιο συνέβη και χθε με την ε, ε, εξυπηρέτηση πεβατών και την Εξυπηρέτηση εδάφου, με συγχωρείτε. Ε, λοιπόν, όσον αφορά τώρα το δικό μας ε, θέμα, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να επιδεινωθεί ποιότητα, δηλαδή τα κριτήρια να κατέβουν προς τα κάτω. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ προτείνω να έχουμε έναν κανονισμό, να καταλήξουμε σε κανονισμό. βεβαίω και μπορούμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα να ρυθμιστούν με την μορφή της επικουρικότητα, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρξουν ενιαίες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, σε αυτό το θέμα θα προχωρήσουμε. Ένα θέμα που θέλω να δείξω είναι παραποίηση. Παραποίηση, πλαστογράφηση ε, των ε, ε, χαρτιών τη άδεια του αυτοκινήτου, του ταχογράφου και πολλών άλλων πιστοποιητικών. Νομίζω ότι οι ε, χώρες ε, οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα προφανώς και επιθυμούν να αφήσουν να ισχύουν και παλιές προδιαγραφές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Η υποτιθέμενη ασφάλεια δεν είναι ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τις, ε, τα δίκυκλα και τις μηχανές, και εγώ εκεί συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν και τους τεχνικούς ε, ελέγχους ε, πράγματι πρέπει να υπάρχει σαφής ε, διαχωρισμός. Δεν μπορεί κανείς να βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα και ένα άλλο καθοριστικό στοιχείο είναι η διάρκεια ζωής, η ηλικία του αυτοκινήτου. Να πω και εγώ για τον εαυτό μου για τα τρακτέρ σύμφωνα με αυτό που ελέγχθη ότι αν έχετε τρακτέρ τα οποία έχουν ρημολκούμενα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση όπως τα φορτηγά. Αν πηγαίνουν όμως από το ένα χωράφι στο άλλο χωράφι δεν έχει νόημα να ελέγχεται ένα τρακτέρ το οποίο κάνει απλώς αγροτικές εργασίες. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και στοχοθετημένοι. Για την τροπολογία του κυρίου Κούν, για την αξιοπιστία των οχημάτων. Λυπάμαι κύριε Κούν αλλά η τροπολογία σας, η 28, είναι ολεθρία για το πώς γίνονται οι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Γιατί όπως είπε ο κύριος ε, Πέρκερ, αν κάποιος αρχίζει να παίζει με το σύστημα, τότε χάνει την άδειά του για να είναι ανεξάρτητο κέντρο ελέγχου. Και υπάρχουν πολλά μικρά συνεργεία και γκαράζ στις στο Ηνωμένο Βασίλειο που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και δεν νομίζω ότι είναι λογική η πρότασή σας και ελπίζω ότι θα επανέφθετε σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει την τροπολογία σας υπαριθμών 5 που μας πιένει στη λάθος κατεύθυνση και έχω και εκεί προβλήματα. Να σας υπενθυμίσω επίσης αυτά που είπε ο κύριος Έλλης στην ακρόαση για τους τροχούς που δεν είναι σωστοί και που πολλές φορές μπαίνουν λάθος ζάντες σε λάθος άξονες. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσετε λοιπόν. Και για τα παρελκόμενα. Εγώ νομίζω ότι τα 1 θα πρέπει να ε, αποκλείονται, ακόμα και τα 0-2 να αποκλείονται από αυτούς τους ελέγχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάρα πολλά μικρά ρημουλκούμενα και δεν πρέπει όλοι αυτοί να πηγαίνουν και να κάνουν κάθε χρόνο ελέγχους για αυτά τα μικρά ε, παρελκόμενα. Να δούμε τα, τα τροχόσπιτα βεβαίως, ναι αυτό έχει νόημα, αλλά τα περισσότερα από αυτά ελέγχονται ούτως ή άλλως και το τελικό μου σημείο. Δεν μπορώ να φανταστώ, ήμουνα σε εμβροντισία όταν είδα ότι υπάρχουν 12 κράτη-μέλη που δεν έχουν τακτικούς ελέγχους στις μοτόρες, στις μοτοσικλέτες. 12 από τα κράτη-μέλη μας, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, δεν ελέγχουν τις μοτοσικλέτες σε τακτικό επίπεδο. Αυτό είναι ε, παράλογο. Κύριο Σοντίδη, από την Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους άλλους οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο για το θέμα αυτό στην Επιτροπή σας. Νομίζω ότι έχετε καταλήξει σε μια σωστή ισορροπία με, σε σχέση με το είδος των ε, ελαχίστων κανόνων που πρέπει να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε αυτό το ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Ξέρω ότι υπάρχει κάποια ευελιξία η οποία εναπόκειται στα κράτη-μέλη για να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές παράμετρους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των οχημάτων μέσα στο οπλοστάσιο ε, εργαλείων που έχουμε για να εξασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια. Προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε μία νομοθεσία που ανατρέχει στο 1977 και έχει μόνο αναθεωρηθεί το 1996. Είναι καιρό να την τροποποιήσουμε για το πώς γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων. Είναι πολύ διαφορετικά τα ίδια τα οχήματα πια σήμερα από ότι τότε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχατε το θάρρος να συνεχίσετε να ζητάτε να υπάρξει συμπερίληψη όλων των οχημάτων και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απάτη στα ταχόμετρα και μας ενδιαφέρει η, και η αντιμετώπιση που προτείνεται για δυνητικά, δυνητικά, δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων στα κέντρα ελέγχου. Και πραγματικά δεν θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν με διαφορετικό τρόπο τους ελέγχους από ό,τι γίνεται σήμερα. Γιατί δεν έχουμε καθόλου στοιχεία που να κατατείνουν στο ότι είτε τα φυσιολογικά ε, γκαράζ ή ένα ειδικευμένο κέντρο μπορεί να είναι καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε κάποιες πρόνοιες που να εξασφαλίσουν τη σωστή κατάρτιση των ε, <clears throat> ελεγκτών και την απουσία σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του επισκευαστή ενός, οχήματο ενός οχήματος και κάποιου που συνδέεται με κάποιο οικονομικό συμφέρον. Για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα, ναι, παρακαλώ, ακολουθήστε τη γραμμή της Κομισιόν και χαίρομαι που αυτό φαίνεται να γίνεται στην έκθεση του κ. Κούν για να συμπεριλάβουμε και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Έχουμε στοιχεία ότι αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας και επίσης υπάρχουν στοιχεία, όπως ε, είπε και ο εισηγητής, ότι τα οχήματα αυτά παρακάμπτουν πολύ σημαντικές πρόνοιες οι οποίες εξασφαλίζουν την οδική ασφάλεια. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα συμφωνούσα και εγώ τα τρακτέρ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σφαίρα εφαρμογή μόνο όταν χρησιμοποιούνται να κάνουν το ίδιο πράγμα όπως ένα εμπορικό όχημα. Όταν κινούνται με υψηλή ταχύτητα στους δρόμους τότε θα πρέπει να ελέγχονται αλλά αυτά τα οποία κάνουν απλώς μια περιστασιακή χρήση των δρόμων για να πάνε στο χωράφι δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τόσο αυστηρές προδιαγραφές. Για τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ναι. Έχουμε δει πολλές προτάσεις οι οποίες βελτιώνουν το κείμενο σημαντικά. Είναι ένας από τους χώρους όπου θα μπορούσε κανείς να απαλύνει τις υποχρεώσεις τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, γιατί για πάρα πολλά κράτη αυτό θα μπορούσε να σημαίνει σημαντικό κόστος και για την πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Και το είδος των κέντρων που χρησιμοποιούνται και τον αυτόματο χαρακτήρα της προσέλευσης των οχημάτων σε αυτά τα κέντρα θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε ένα πιο ευέλικτο τρόπο τουλάχιστον μεταβατικέ διατάξεις για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν. Για τις νομικές πλευρές. Είναι σημαντικός ένας κανονισμός και χαιρόμαστε που ο εισηγητής θέλει να διατηρήσει αυτή τη ρύθμιση. Δεν στρέφεται κάτι σαν αναλογικότητος. Ο κανονισμός μας δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύπτονται και πολλά τρίτη μέρη από υποχρεώσεις. Τέλος ε, λοιπόν όσον ε, αφορά στην ε, ετήσια, στον ετήσιο έλεγχο των οχημάτων, εδώ αυτή είναι η μόνη απογοήτευση από δική μας πλευράς. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αρκούν ε, για να αποδείξουν ότι θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα ε, οχήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον όσον αφορά τον ε, αριθμό των ε, χιλιόμετρων. Και το γεγονός ότι σαγάγαμε τα 160.000 χιλιόμετρα, αυτό δεν το βρήκαμε από το μυαλό μας, απλά διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει ένα κριτήριο και αυτό ήταν το πιο αντικειμενικό κριτήριο έτσι ώστε από αυτό τον αριθμό χιλιόμετρων και μετά τα ε, οχήματα να ελέγχονται σε αιτήσια βάση. Τα αποδεκτικά λοιπόν στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα και νομίζω ότι υπάρχει και ε, κάποια δυνατότητα να εφαρμόζονται περιβαλλοντικές προδιαγραφές γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να αποδείξει ότι πρέπει και μπορούν να βαθμιστούν όλα τα αυτοκίνητα έτσι ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, κύριε Σιγητά, θέλετε να πείτε κάτι, ε, αλλιώς θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για ένα θέμα, δηλαδή για το ότι ε, μπορούμε να επιβάλλουμε τις ε, τεχνικές ε, προδιαγραφές. Βεβαίως διαφωνούμε όσον αφορά τους ελεγκτές, ε, κατά πόσον θα πρέπει να είναι επιστοποιημένα συνεργεία ή ανεξάρτητες μονάδες, αλλά το να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, αυτό είναι σημαντικό. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο και σε ένα πιστοποιημένο συνεργείο. Ε, τώρα, όσον αφορά τα τρακτέρ, ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά δουλεύουν στα, ε, στους αγρούς και μετά, εντάξει, κάνουν και ένα μικρό διάστημα στην άσφαλτο. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να ελέγχονται απαραίτητα. Αλλά τα άλλα τρακτέρ τα οποία μεταφέρουν ε, τα σιτηρά ας πούμε, και διανύουν αποστάσεις 60-70 χιλιόμετρων, αυτά θα πρέπει να ελέγχονται. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο των δίκυκλων, νομίζω ότι σχετικά με αυτό θα βρούμε κάποια λύση και ε, απευθύνομαι σε όλους, σε, σε όλους εκείνους που είπαν ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε και να δίνουμε άδεια σε μηχανές ε, που τρέχουν με πάνω από 300 χιλιόμετρα στα ιστορικά αυτοκίνητα και εκεί συμφωνούμε ε, πράγματι και κάποιες ε, μοτοσικλέτες δεν χρειάζεται να ελέγχονται, εξαιρούνται. Νομίζω λοιπόν ότι ορισμένα πράγματα μπορούμε να τα διευκρινίσουμε. Και όσον αφορά τα ρημουλκούμενα οχήματα, ας καθορίσουν τα κράτη-μέλη πώς θα ορίζουν τα ρημουλκούμενα οχήματα. Και όσον αφορά την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αυτή τη βρίσκω πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, να έχουμε στο, διαβατήριο, στο αυτοκίνητο ένα διαβατήριο που να περιγράφονται όλα τα τεχνικά του στοιχεία. Αυτό θα επιφέρει διαφάνεια και λιγότερες ε, αντιπαραθέσεις. Και χαίρομαι ε, για την ε, συνεργασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολλά από τα θέματα απαντήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλοί και καλοί λόγοι να ελέγχουμε τα εμπορικά οχήματα 3,5 τόνων. Είναι μια κατηγορία που πρέπει να μας απασχολεί. Τώρα το 5% απαιτεί παρετέρω συζήτηση. Πάντως, η πρόταση του κύριου Φέρμπερ μου φάνηκε ενδιαφέρουσα να εισάγουμε δηλαδή ένα νέο σύστημα υπολογισμού του ποσοστού αυτού. Αλλά θα έπρεπε το νούμερο να το αποφασίσουμε μετά από μια μελέτη που θα γίνει για τα ελαφρά οχήματα, ώστε να δούμε τελικά ποιε θα είναι οι επιπτώσει. Ένα σύστημα τώρα εκτίμηση κινδύνου επίση είναι κάτι που θέλω να υποστηρίξω, γιατί δεν πρόκειται για επιθεωρήσεις για την επιθεώρηση, έλεγχη για τον έλεγχο, όχι, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο και έχουμε εμπειρίες από το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ άλλων που δείχνουν ότι το θέμα δεν είναι η τιμωρία. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανένα, να επιβάλλουμε κυρώσει σε μια επιχείρηση, σε οποιοδήποτε άλλον. Δεν πρόκειται για την επιθυμία μας να κάνουμε έλεγχο για τον έλεγχο. Έπειτα, η ασφάλεια του φορτίου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Τώρα θέλω πώς πω κυρία Γκρίσπερκ για την τροπολογία αριθμός 5. Εκεί ακριβώς θέλουμε να αντικατοπτρίζεται και η ιδέα της ε, διαφοροποίησεις της χιλιομετρικής απόστασης, το 10 χιλιόμετρων δηλαδή. Όταν μιλάμε για σημεία ε, όπου υπάρχουν κέντρα ελέγχου και αυτά πρέπει να βρίσκονται στην γύρω περιοχή, γι' αυτό το αφήνουμε έτσι και δεν βάζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Η εναρμόνιση και γιατί πρέπει να γίνει, ε, νομίζω ότι είναι σαφές και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να γίνει και κανονισμός. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πρώτα απ' όλα, δεν συμφωνώ για τις προθεσμίες όσον αφορά τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Αν έχουμε μεγάλη προθεσμία, τότε η πρόοδος θα προχωρήσει πολύ αργά και εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το μέλλον. Όσον αφορά την κυρία Τικάου, αλλά έφυγε δυστυχώς από ό,τι βλέπω, θα έλεγα ότι καιρό εγώ κάθισα και σκέφτηκα πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντα μπορούμε να εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη ενός οχήματος. Ίσως μπορούμε να αλλάξουμε κάπως τη διατύπωση. Αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία Τικάου κατάλαβε τι εννοώ εγώ με την τροπολογία που έχω καταθέσει. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ωραία προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 25 Μαρτίου, ε, 27 Μαρτίου τροπολογίες που στις 22 και 23 Απριλίου θα εξετάσει η Επιτροπή μας και θα ψηφίσουμε εδώ 30 Μαΐου. Οπότε πρώτος στόχος 27 Μαρτίου υποβολή κατάθεσης ε, τροπολογιών. Εδώ έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών του κύριου Κράμερ. Καλώς ήρθατε. Και λυπάμαι που πρέπει να είσαστε όρθιοι και να μην μπορείτε να ακούσετε και τη διερμηνία έτσι ώστε να καταλάβετε τι συζητάμε. Η δίκηση, βλέπετε, του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι αυτή είναι μια εξαίρετη αίθουσα για τις συνεδριάσεις μας. Εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια. Δεν συνεδριάζουμε πάντα εδώ και τυχαίνει σήμερα να μας πετυχαίνετε στην χειρότερη κατάσταση ποτέ, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Δεν θα μπορούσα να καθίσω στις κενές θέσεις. Γιατί όχι, υπάρχουν και νέες θέσεις, δεν μπορούν. Δεν ξέρω, η δικιά μου η εμπειρία είναι ότι άπαξ και πάει και καθίσει κάποιος σε μια καρέκλα που δεν δικαιούται, ορμάνε και τον ε, σηκώνουνε. Καλά, εντάξει, εγώ το είπα γιατί θεώρησα ότι θα ήταν μια λύση. Πρόεδρος, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας, αλλά τέλος πάντων. Επόμενη έκθεση έκθεση του κ. Higgins για τα τηλεδιώδια, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θυμόσαστε ότι σε μια προηγούμενη συνεδρία είχα δώσει μια σύντομη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Για να σας υπενθυμίσω, εδώ και πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει τις οχλήσεις στη διέλευση των συνόρων να έχουμε μια ενιαία αγορά χωρίς ε, ε, φραγμούς. Και ένα τέτοιο στοιχείο για τις μεταφορές είναι να μην υπάρχει κάποια στρέβλωση λόγω των τελών και διακρίσεων κατά οχημάτων. Από την άλλη μεριά να υπάρχει ε, προτιμησιακή μεταχείριση για τα λιγότερα ρηπαίνοντα οχήματα. Επίσης πρέπει να, να εξασφαλίσουμε ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της οδική υποδομής. Πώ μπορούμε λοιπόν να προωθούμε την οδική υποδομή και να καταλογίσουμε το κόστο της με δίκαιο τρόπο, χωρίς να παραδιάσουμε τις τέσσερι ελευθερίε της ενία αγοράς. Και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει την χάνει σεβασμού. Και τέλο ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο, να εφαρμόσουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα τηλεδιοδιών, το EETS όπως το λέμε στα Ιρλανδικά. Αυτό είναι λοιπόν ο στόχος της έκθεσής μου. Η Κομισιόν έχει εκδώσει δύο ανακοινώσεις, μία για την ε, επιβολή τελών από ελαφρά οχήματα και το δεύτερο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τηλεδιοδιών, το EETS. Είναι συνδεόμενα θέματα που έχουν να κάνουν με τον καταλογισμό τελών στους δρόμους. Κάθε μία από τις δύο προτάσεις όμως έχει διαφορετική εστίαση και η έκθεση αυτή που έχετε ενώπιόν σας βασίζεται σε αυτές τις δύο ανακοινώσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε αναλογικό καταλογισμό τελών. Τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν ένα σύστημα επί βάση χρόνου θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Αλλά τα τέλη θα πρέπει να έχουν αναλογικό χαρακτήρα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να έχουν καταλογισμό σε ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο καταλογισμό κτλ και θα πρέπει εκτός από το διοικητικό τέλος να είναι αντίστοιχα με αυτά που έχει κανείς για μια βινιέτα η οποία θα πρέπει να είναι αναλογική ας πούμε γιατί χρήση της εβδομαδία κτλ. Αυτή τη στιγμή σε κάποια κράτη-μέλη η εβδοματία βινιέτα μπορεί να είναι μέχρι τέσσερις φορές σε αναλογικό επίπεδο το κόστος μιας ετήσιας βινιέτας και αυτό για πολλούς θεωρείται ότι είναι ε, άδικο για οχήματα που δεν προέρχονται από αυτό το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Και σε ό,τι αφορά τις βινιέτες, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα για να καταλογίσουν το κόστος χρήσης των υποδομών τους, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και σαφέστερες διασφαλίσεις και προορίες ώστε κρατη μέλη να μπορούν να καταλογίζουν κόστος επί τη βάση προορατά αναλογικά, συν ένα μικρό διοικητικό τέλος. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει ως το πιο απλή η χρήση αυτών των βινιετών και πώς τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να κάνουν αυτό και όχι να καταλογίσουν με άλλους τρόπους τα τέλη. Η Κομισιόν έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή και συνόρμηση και τη δυνατότητα να μπορούν να αγοράζουν με εύκολο τρόπο οι αυτοκινησιστές της βινιέτες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και τη δυνατότητα να πληροφορήσουμε καλύτερα τους ε, οδηγούς πώς καταλογίζεται το κόστος της βινιέτας και για το περιβάλλον. Είναι ο καταλογισμός τελών ένα σημαντικό τρόπο για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή τη αρχή ο πληρώνων ρηπαίνει κιόλα. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη για ρυθμίσει για τα ευρωτηλεδιώδια. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν είναι απλό αυτό το θέμα και η Κομισιόν δεν έχει πράξει αρκετά για να εξασφαλίσει ότι τα ευρωτηλεδιώδια γίνονται μια πραγματικότητα. Ελπίζω ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορέσουν να συμμετάσχουν για να γίνει πιο ρεαλιστικό αυτό το σχήμα και αυτή τη στιγμή βέβαια δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για την κατεύθυνση αυτή. Ε, τα τέλη για όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να γίνουν μια πραγματικότητα για όλους στο ορατό μέλλον. Θα πρέπει τα αυτοκίνητα να είναι πιο αποτελεσματικά στη χρήση των καυσίμων και, και η επιβολή τελών για την χρήση των δρόμων θα πρέπει να επαφείται στα κατημέλη, αλλά με την υποχρέωση να είναι αναλογική αυτή η επιβολή. Με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει ένα κανονισμό για τη χρήση των υποδομών για να μπορούν να συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις τη Ευρωπαϊκή Υποδομή Δρόμων στο μέλλον με τη χρήση διοδίων. Και φαίνεται ότι οι κατευθυντέ αυτές γραμμές είναι επαρκείς για τις βινιέτες. Και καταλαβαίνω ότι πολλά κράτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τύχη πιέσεων από λόμπι όπως είναι εθιμικά ε, εύλογο για τέτοια θέματα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει αγορά για τα ευρωτηλεδιώδια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι εφικτή αυτή η ρύθμιση, αλλά δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά οι ιδιωτικέ εταιρείε από την διαλειτουργικότητα και κάποιες εταιρείε μπορεί ακόμα να χάσουν και τα κέρδη τους. Αλλά αυτός δεν είναι από χρόν λόγος να απορρίψουμε την εφαρμογή του EETS, το οποίο είναι ανοιχτό σε όλους και δεν έχει φραγμούς για κανένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Mr. Higgins. Mrs. Meissner. Ευχαριστώ, κύριε Meissner. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω Α, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χικίν για όλα αυτά που μας είπε και θέλω να σας πω ότι τώρα δεν ομιλώ εξ ονόματός μου, αλλά εξ ονόματος του κυρίου Κλίν, σε του σκιώδους εισηγητού μας, ο οποίος όμως μου εξέφρασε τις απόψεις του και λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να αποφασίζουν, μόνο τους αποφασίσουν, τι θα κάνουν σχετικά με τα διόδια. Λέει, ας πούμε, στη Ρουμανία το ύψο των διοδίων δεν μπορεί να είναι το ίδιο όπως στη Γαλλία και δεν πρέπει να είναι. Άρα δηλαδή ε, το ύψο των να παραμένει στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Να υπάρχουν επίσης διαφανείς μηχανισμοί ε, κυρίως όσον αφορά την επιβολή κόστους. Ε, ο μηχανισμός ε, πληρωμής να είναι πάρα πολύ απλός και να μπορεί κανείς και πολύ εύκολα να αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατά τα άλλα, ο κύριος Κλίνς ε, χαιρετίζει το γεγονός ότι το όλο θέμα τον έλαβε ο κ. Χίκινς ε, να μπορεί κανείς να αγοράσει αυτοκόλλητα σήματα στο μέλλον ηλεκτρονικά. Αυτό οπωσδήποτε είναι φιλικό προς το περιβάλλον και εύχριστο. Επίσης, σωστά λέει ο κ. Χίκινς, ε, να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σήμα που να δείχνει ποιες διαδρομές υπόκεινται σε διόδια και ποιες όχι. Ας πούμε, εγώ στην Αυστραλία που είχα πάει δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς ε, ενημερωμένος ε, και να γνωρίζουν οι καταναλωτές. Τώρα, είτε διόδια είτε αυτοκόλλητα σήματα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της κοινή αγοράς που είναι ελεύθερη μετακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων, ε, κεφαλαίου. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δίδεται σημασία στην διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Επίσης, δεν επιθυμούμε να υπάρχει διακριτική μεταχείριση των χρηστών ε, λόγω εθνοτικής προέλευσης ή ε, παραμονής μόνιμης εγκατάστασης, χώρου μόνιμης εγκατάστασης. Να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση. Ο κύριος Εγκίνης λέει ότι θα πρέπει στην αγορά να εμφανιστούν καινούργοι πάροχοι. Κατά τα άλλα, ε, χαίρεται και προσβλέψει διαπραγματεύσει και την επόμενη φορά θα είναι οπωσδήποτε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γιάλα Σέντερ, τη σκιώδη ηγετριά μας, δεν μπορεί να είναι εδώ τώρα. Οπότε εγώ την αντικαθιστώ και θα διαβάσω την άποψή της στα αγγλικά, επιτρέψτε μου. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες ε, κάποιων ε, φορέων που εποφολούνται λίγο από την Ευρωπαϊκή Ευθυπηρεσία Τηλεδιοδίων, όμως δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Πάρα πολλές χώρες ε, υποφέρουν από την αδυναμία να έχουν πρόσβαση στην καρδιά της ευρωπαϊκής ε, αγορές. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με προτάσεις οι οποίες να επιταχύνουν την διαδικασία. Φοβούμεθα ότι αν αφήσουμε αυτή τη διαδικασία στους φορείς δεν θα υπάρξουν πλεονεκτήματα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δει τι κίνητρα μπορεί να υπάρχουν και να λύσει ό,τι προβλήματα προκύπτουν. Προς το παρόν ε, μπορούν ε, τα φορτηγά να προχωρούν και να περνάνε από διάφορες χώρες με ενίες μεθόδους. Υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ δύο χωρών για τα φορτηγά. Θα έπρεπε να υπάρχει και για άλλα οχήματα όπως ε, συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό θα έπρεπε να είναι εφικτό και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χαιρόμαστε για την ε, πρόταση του εισηγητή για να χρησιμοποιηθούν διάφορα δορυφορικά συστήματα, μια που έχουν ήδη γίνει σχετικές επενδύσεις, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν παρετέρω. Τέλος, Όσον αφορά την χρέωση, εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να λυθεί περισσότερο η λύση χρέωσης βάση απόστασης και όχι βάση χρόνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χίγγιν, τον εισηγητή. Έχω κάποια σημεία που θέλω να θίξω. Φυσικά αυτό που είναι σημαντικό είναι να αναγνωρίζει η έκθεση ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα να αποφασίζουν για το ύψος των ε, τελών και να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν και τα έσοδα από τη χρέωση αυτή. Τώρα, όσον αφορά την διαλειτουργικότητα, όντω το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να έχει την διαλειτουργικότητα. Αλλά Άπαξ και υπάρχουν ρυθμίσεις, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει κάποια ισορροπία σύμφωνα με την ε, χρήση του δρόμου. Ορισμένοι μπορεί να μην επωφελούνται από την διαλειτουργικότητα γιατί αυτό τους ε, επιβάλλει παραπάνω έξοδα, ιδιαίτερα εάν δεν ε, κυκλοφορούν σε πολλές χώρες συγχρόνως. Εγώ, ας πω, έρχομαι από ένα νησί, ένα τέτοιο σύστημα δεν θα μας ευνοούσε. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Υπάρχει ήδη πάντως οδηγία για να καθοριστεί πλαίσιο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων. Πρέπει να διευκρινιστεί τι τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί. Κάποιες χώρες τη χρησιμοποιούν. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα της χρέωσης. Η δικιά μου χώρα και φαντάζομαι κι άλλες. Εντάξει, πολλά επιχειρήματα ακούγονται για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνεται η χρέωση βάση απόστασης ή βάση χρόνου. Προς το παρόν έχουμε το σύστημα της βινιέτας του αυτοκόλλητου σήματος. Θα πρέπει να δούμε και τα άλλα συστήματα. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιστραφεί η διαδικασία που ισχύει σήμερα. Ευχαριστώ τον Τζιμ πάντως. πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να προχωρήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις βέβαια όλων των χωρών. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Καντσίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε και κύριε Higgins ε, για το έγγραφο που καταθέσατε και έρχεται σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Κοιτάξτε, αυτά που θέλω να πω θα τα πλουστέψω. Τέσσερα είναι βασικά τα σημεία. Σημαντική λοιπόν καταρχήν είναι η διαλειτουργικότητα των μέσων. Προφανώς και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης ε, είναι σημαντικό να είναι κανείς ενημερωμένος σχετικά με το κόστος. Γιατί από τη στιγμή που εντάσσομαι σε ένα ε, δορυφορικό ε, σύστημα ενδέχεται στο τέλος να έχω να αντιμετωπίσω κάποιο κόστος το οποίο όμως δεν γνωρίζω ευθύς εξ αρχής. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Και τέλος, ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος ε, χωρίς ειδικούς φραγμούς. Αυτός είναι σημαντικός στόχος που έχει βέβαια άμεση σχέση με την ιδιωτικότητα γιατί σήμερα υπάρχουν αυτά τα συστήματα τα free pass που έχουν άμεση σχέση με την δορυφορική πλοήγηση, αλλά όταν μπαίνει κανείς στην δορυφορική πλοήγηση θα πρέπει να έχει πάντα κατά νου την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Τα άλλα συστήματα που υφίστανται, ε, τα άλλα αυτά συστήματα ε, έχουν κάποιους φυσικούς φραγμούς και δημιουργούν προβλήματα. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν μιλάμε για ποσά, αλλά μιλάμε για συστήματα. Στις διάφορες χώρες ε, υπάρχουν και διάφοροι πάροχοι για διαφορετικά συστήματα υπάρχουν ε, συστήματα ιδιωτικά και δημόσια. Εγώ βέβαια δεν γνωρίζω κατά πόσο ο κανονισμός είναι η σωστή λύση λόγω του ότι, όπως σας είπα, υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ε, το GPS ε, να αποκαλείται GNSS, η κατάσταση αυτού του αρκτικόληξου, επ' αυτού συμφωνώ και στο σημείο υπαριθμών 3 πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, προσθέσουμε το εξής, ότι όποιος ε, προσφέρει την υποδομή θα πρέπει να προσφέρει και τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν την υποδομή. Να προσθεθεί δηλαδή αυτό το τελευταίο. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι είναι ευκταίο τα κονδύλια να επανέρχονται στον τομέα των ε, μεταφορών έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να ε, τροφοδοτείται και η, η τεχνολογία που είναι απαραίτητη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να έχουμε πάντα κατά νου και τις διαδρομές, τις αποστάσεις αλλά και τη ρήπανση. Αυτές τις προσθήκες έχω, έχω να κάνω και εύχομαι ε, στο Jim να συνεχίσει την πάρα πολύ καλή δουλειά που μας παρουσίασε μέχρι σήμερα. Ο κύριος Χέντμπερκ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή τον κύριο Χίγγενς για την έγκαιρη έκθεση του. Η Κομισιόν σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί με τη διάγνωση του εισηγητή ίσως όχι όμως και με όλες τις συνταγές. Δύο ή τρία σημεία στα γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα διόδια και τα τέλη. Ιδίω για τα βαρέα αυτοκίνητα, καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν θα μπορούσε φέτος να προχωρήσει σε μια προ βουλία για να υπάρχουν τέλη βάση αποστάσεως που διανύεται. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό και δίκαιο για την καταβολή τελών και ιδίως να εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών εθνικών συστημάτων και ίσως να υπάρξουν και πρόνοιες για τα επιβατικά αυτοκίνητα που να αφορούν την συμφόρηση στις πόλεις, την ε, <clears throat> διαφοροποίηση της χρήσης τους και σε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση τα κύρια κίνητρα θα ήταν να εξασφαλίσουμε για τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο, το αυξανόμενο ε, δημοσιονομικό χάσμα μεταξύ των εσόδων και της, του κόστους των, της οδικής υποδομής που είναι πρόβλημα για όλες τις χώρες και δεύτερον να μπορέσουν πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν τη συμφόρηση που γίνεται μια όλο και μεγαλύτερη πρόκληση με συνεπακόλουθο οικονομικό κόστος, γιατί είναι πραγματικά απώλεια εσόδων σε οικονομικό επίπεδο. 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνεται, 1% του παραγωγικού ΑΕΠ, γιατί χάνεται ε, χρόνος εργασίας, χάνεται βιομηχανικό και η παραγωγή που βασίζεται σε έγκαιρες παραδόσεις κτλ. Τώρα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τηλεδιοδίων. Η Κομισιόν έχει προωθήσει ενεργά τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Πιστεύουμε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο για ένα τέτοιο σύστημα έχει πράγματι εφαρμογή στην, ε, ακολουθώντας τη γαλλική ε, πρόταση για το οικολογικό ε, φόρο για τα φόρτηγα. Η Επιτροπή Αρμόδια για τα Διόδια έχει συναντηθεί τέσσερις φορές και έχει πάρει το Κοινοβούλιο μία έκθεση για τις συναντήσεις αυτές. Αν τώρα δεν επιτευχθεί επαρκής πρόοδος για την εφαρμογή του EETS του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τηλεοδίων, με ένα κατάλληλο σχήμα. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να προτείνει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες εάν χρειάζεται. Και επίσης αναφέρθηκε από ορισμένου βουλευτές ότι υπάρχουν τέσσερις κατασκευαστές ε, εξοπλισμού που έχουν αναπτύξει ε, εξοπλισμό για τα φορτηγά που να είναι συμβατός και με το γαλλικό σύστημα ECOTAX και με το EETS. Και υπάρχουν έξι εταιρείε οι οποίες λένε ότι μπορούν να καλύψουν με ένα μονάχα, με μία συσκευή μονάχα, Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την καταληκτική ημερομηνία του Οκτωβρίου του 2012 για τα βαρέα αυτοκίνητα, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε απόρριψη του βρέφους μαζί με τα ύδατα κολύμβησης του ίδιου αυτού βρέφους. Το σύστημα αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται από 7 κράτη-μέλη που έχουν ε, σημαντικά συστήματα διαιωδίων και μεγάλη κάλυψη σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των φορτηγών. Εμείς λοιπόν ακόμα διατηρούμε το φέλημα της αμφιβολίας για τα θέματα αυτά και πιστεύουμε ότι τον τρόπο αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε ιδιαίτερα σε μια έγκαιρη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τηλεοδιοδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν βλέπουμε πώς αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος, αλλά εάν δεν είναι ικανοποιητικό, η Κομισιόν θα εξετάσει και άλλες επιλογές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χίγγινς, θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά. Όχι, Πρόεδρε. Απλώς τρία λεπτά. Νομίζω ότι υπάρχει γενική υποστήριξη για την κύρια κατεύθυνση της έκθεσης. Θέλω ευχαριστώ κυρία Μάσνα και την κυρία Φώστερ και ο κύριος Κιάν Κέν είχαν ακριβώς το ίδιο επιχείρημα ότι τα κράτη θα πρέπει να αποφασίσουν για το κόστος των τηλεδιοδιών. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που θα είναι σαφής και διάφανος. Το να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύμβολο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε ένα αναγνωρίσιμο σύμβολο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όσα έχουν. Υπάρχει τεχνολογία. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η πολιτική θέληση και νομίζω ότι ότι μία αντιμετώπιση που να βασίζεται μόνο στην απόσταση είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε. Για αυτά που είπε η κυρία Φώστερ. Υπάρχει το θέμα της διαλειτουργικότητας από ένα κράτος στο άλλο. Υπάρχουν κράτη τα οποία βασίζονται σε εξαγωγές όπως είναι η Ιρλανδία και επομένως τα φορτηγά μας κυκλοφορούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είναι νευραλικό το θέμα για μας. Για το κόστος ο κύριος Κάνκεν τόνισε Μα εδώ δεν θέλουμε να θεσπίσουμε ένα νέο σύστημα. Υπάρχει τεχνολογία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε λειτουργική και διαλειτουργική αυτή η τεχνολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρησιμοποιούμε νέε τεχνολογίε λοιπόν και γι' αυτό οι εταιρείε δεν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο γιατί δεν πρόκειται να βγάλουν πρόσθετα λεφτά. Αυτό το οποίο χρειάζεται τελική ανάλυση είναι η πολιτική θέληση για να λειτουργήσει αυτό. Και για αυτά που είπε η Κομισιόν καταγράφω αυτά που λένε, αναφέρθηκαν και στο κόστος συντήρησης τη οδικής υποδομή στην Ευρώπη που γυράσκει. Επίσης τα θέματα της συμφόρησης στου δρόμου. αυτό είναι απώλεια 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και για την περιφερικοποίηση ξέρω ότι αυτό το οποίο ε, επεξεργάζεστε απαιτεί μια κρίσιμη μάζα αν βρείτε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ότι η περιφερικοποίηση δεν λειτουργεί, ελπίζω ότι θα προχωρήσετε με μια νομοθετική πρόταση και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο. Και... Και εμεί σα ευχαριστούμε κύριε Higgins. Η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών 25 Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι υποθέτω και η ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή θα γίνει στις 23 Απριλίου. 25 Μαρτίου το μεσημέρι είναι η διορία για την κατάθεση των τροπολογιών. Ε, τώρα πάμε στο επόμενο θέμα σχετικά με τις, ε, τους τριμερείς διαλόγους. Και θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω. Μετά ε, θα μιλήσουν οι υπόλοιποι και ο κύριος Κουμουτσάκος Είχαμε λοιπόν τρεις ε, συναντήσεις. Η έλαβε χώρα στις 27 Φεβρουαρίου, όπου ο κύριος Κουμουτσάκος και η κυρία Μάισνερ παρίσταντο. Ε, νομίζω ότι ε, σημειώσαμε πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές διαφορές όσον αφορά το θέμα των ρητρών non-regression και no ratification. το θέμα είναι κατά πόσον τα δικαιώματα των ...αυτεργατών θα πρέπει να προσθεθούν στα παραρτήματα. Ε, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και ε, βεβαίως ε, το θέμα της, του κράτους σημαίας αυτό είναι θέμα της Επιτροπής. Μήπως έχει κανείς ερωτήσει από αυτού. Αν όχι, πάμε στα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα. Γιώργο, θες να ξεκινήσεις. Είχαμε τον πρώτο τρίλογο στις 20 Φεβρουαρίου. Έχουν ε, προβλεφθεί ακόμα τρεις. Ο επόμενος είναι στις 21 ε, Μαρτίου, δηλαδή μεθαύριο ο επόμενος τον Απρίλιο και ο τελευταίος ε, τον Μάιο. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμα ένας, ακόμα μια συνάντηση πέραν εκείνης που προβλέπεται ως καταληκτική αυτή τη στιγμή για τον Μάιο. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν ακόμα μία. Πρέπει να πω ότι το κλίμα ήταν θετικό. Η εντύπωση που αποκομίσαμε από τον τρόπο που η Ιρλανδική Προεδρία σκοπεύει να χειριστεί το θέμα Νομίζω ότι η εντύπωση είναι ότι θα υπάρξει μια σχετική ευελιξία και καλή πρόθεση εκ μέρους της. Αποφασίσαμε σε αυτή την ε, συνάντηση επίσης ορισμένα μεθοδολογικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Τρίλογος. Πρώτο βήμα, ότι καλό είναι οι συναντήσεις του Τριλόγου να προετοιμάζονται σε τεχνικό επίπεδο από πριν, ώστε οι συζητήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικές όταν φτάνουμε στο επίπεδο του τριλόγου. Έχουν γίνει ήδη δύο τέτοιες τεχνικού επίπεδου συναντήσεις. Το δεύτερο μεθοδολογικό, η δεύτερη απόφαση για τη μεθοδολογία ήταν να προσεγγίσουμε το κείμενο σε θεματικές ομάδες και όχι άρθρο προς άρθρο είτε κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα για ένα θέμα το οποίο είναι διασπασμένο μέσα στο κείμενο να κάνουμε μια συνολική και σφαιρική συζήτηση. Κατά την ε, πρώτη αυτή συνάντηση είχαμε επίσης την ευκαιρία και από πλευράς Κοινοβουλίου αλλά και το Συμβούλιο μετά να συμφωνήσουμε σε δύο βασικές έννοιες που διατρέχουν όλη τη συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πρώτον, στην αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ως προς τον ορισμό που έχουμε εντάξει στο δικό μας χαρτί, αλλά η βασική θεματική έννοια, η βασική αρχή της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας είναι σεβαστή και από το Συμβούλιο και η δεύτερη θεμελιώδης αρχή που και το Συμβούλιο αποδέχθηκε είναι ότι η μεθοδολογία δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια των τριλόγων. Όσον αφορά, ε, επίσης είχα την ευκαιρία να θέσω προς το Συμβούλιο την δυσαρέσκεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξέλιξη της συζήτηση για τις ε, ε, Multinational Financial Framework. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νέα είναι αρνητικά από αυτό, σε αυτό το επίπεδο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και είχα την ευκαιρία να το θέσω προς το Συμβούλιο χωρίς να πάρω πρέπει να σας πω μια αρκετά πιστική απάντηση. Ε, όσον αφορά τα άλλα ζητήματα, η συζήτηση εστιάστηκε περισσότερο στο άρθρο 4 που έχει να κάνει με τους διαδρόμους, τις πλατφόρμες διαδρόμων και τους συντονιστές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό θα σας αναφέρει ο συνάδελφος κύριος ε, Ερτούγκ θεωρώ ότι είναι θετικό ότι από πλευράς Ελλαδικής Προεδρίας φάνηκε να γίνεται αποδεκτό εκ μέρους, της, εκ μέρους η αρχή των implementing decisions. Τέλος, συζητήσαμε και για τους χάρτες. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει αν οι τροπολογίες που είχε επιφέρει το Συμβούλιο στους χάρτες είναι σύμφωνες οι τροπολογίες αυτές με τη μεθοδολογία, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Έτσι μπορεί να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες του Συμβουλίου, όπως δεκτές οι τροπολογίες που έχει καταθέσει επί των χαρτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μεγάλο βαθμό έχουν γίνει, ε, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, έχουν γίνει δεκτές και από το Συμβούλιο. Είναι βέβαιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ε, στο στάδιο αυτό στις θέσεις του. Ε, αυτός νομίζω ήταν ο άξονας και το περίγραμμα της πρώτης συζήτησης του Τριλόγου ε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα έχουμε, τις ευκαιρίες, θα έχουμε ευκαιρίες να ε, σας ενημερώνουμε για κάθε βήμα και για την πορεία αυτής της όχι εύκολης αλλά πολύπλοκης διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Ερτούκ θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στα επιμέρους ζητήματα που συζητήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ja, vielen Dank, <clears throat> Herr Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γιώργο για τα θέματα περιεχομένου που έχουμε ήδη αντιμετωπίσει για πρώτη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγητές γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ενωτικά και είναι πολύ καλό το θέμα αυτό, το σημείο αυτό. Όπως ανέφερε ο κύριος Κουμουτσάκος, στις 22 Φεβρουαρίου συναντηθήκαμε και την Πέμπτη θα κάνουμε τον δεύτερο, τη δεύτερη συνάντηση τριμερούς διαλόγου. Εμείς από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε δώσει μία ε, σαφή θέση την οποία έχουμε κάνει σαφή και στο Συμβούλιο ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αν θέλουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε κάποια μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό πρέπει να το έχουμε και από την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει αυτό. Επίση, η προσέγγιση επί τη βάση διαδρόμων είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλουμε επίση να υπάρξει και μια πιο ενιαία αντιμετώπιση τη ανάλυση κοινωνικού και οικονομικού ε, κόστου σε σχέση με την ωφέλεια. Είναι κάτι επίση το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει με μεγάλη πλειοψηφία ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής καθορισμός των στόχων ώστε με τα λίγα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα στα TNT να μπορέσουμε τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε προκρίνει να τα χρηματοδοτήσουμε. Επίσης έχουμε τονίσει την ανάγκη να υπάρξουν δεσμευτικά ε, χρονικά όρια και να μην υπάρξει και περιορισμός σε σχέση και επιφυλάξει σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της, ε, μεταξύ της ανάπτυξης των εσωτερικών, της ανάπτυξης των εσωτερικών υδατήρων δρόμων και των οδικών αξώνων και συνδρομικών αξώνων. Πρέπει να βρούμε τη σωστή λοιπόν ε, ισορροπία που θα εξασφαλίσει και την μεγαλύτερη βιωσιμότητα και αηφορία στο μέλλον. Μπορείτε να <clears throat> φανταστείτε επίσης ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων, αλλά αυτές θα αποκρισταλωθούν και σε επόμενες εβδομάδες και γι' αυτό είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλοι και να έχουμε ένα κοινό ορισμό του τι αποτελεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη θέση και επίσης τα κονδύλια του TNT θα πρέπει να αποδοθούν για τη χρηματοδότηση σχεδίων που καταδεικνύουν μια πραγματική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και όχι μονάχα την εθνική προσθέμενη αξία που έχουν τα κρατημέλη πολλές φορές στο μυαλό τους. Και επίσης, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, πρέπει να αναφερθώ και στο θέμα της ε, διαπραγμάτευσης του πολιετούς πλαισίου και αυτό περιλαμβάνει και την, ε, το σχέδιο Connecting Europe. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά. Εδώ πέρα δεν μπορεί να περικόπτει το Συμβούλιο χρήματα και από την άλλη πλευρά να νομίζει ότι μπορούν να συνεχίσουν όλα αυτά τα προγράμματα χωρίς να αλλάξει τίποτα. Επομένως, θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσει ότι είναι απαραίτητο να διαλέξει και το Συμβούλιο ποια σχέδια θα χρειαστεί να διαγραφούν εν ανάγκη. Ο στόχος μας είναι να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρχει και απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόσθετο γραφειοκρατικό άχθος στα σχέδια αυτά. Και αυτό ιδιαίτερα αφορά το κεφάλαιο 4 για τους διαδρόμους. Το Συμβούλιο επίσης θέλει να περιορίσει το ρόλο του συντονιστή. Μπορούμε να φανταστούμε γιατί. Για να υπάρχει ώστε να τον μικρότερη παρέμβαση και επιρροή από την πλευρά της ευρωπαϊκής διάστασης, αυτό το οποίο φυσικά εμείς απορρίψαμε. Και επίσης το Συμβούλιο δεν θέλει να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το συνολικό δίκτυο. Εμείς έχουμε θέσει σαν χρονικό οριζόντα το 2050 και επίσης το Συμβούλιο δεν φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα για ένα σαφή ορισμό της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Τέλος, το Συμβούλιο θέλει να έχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα να καθορίζει τις εξαιρέσεις και τους τεχνικούς κανόνες σε ορισμένα σημεία. Στον πρώτο τριγωνικό διάλογο καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι πολλές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορούν να γίνουν αποδεκτές, να εντοπιστούν τουλάχιστον, να ταυτοποιηθούν αυτές οι τροπολογίες που μπορεί να είναι αποδεκτές για το Συμβούλιο και έτσι οι τεχνικές συναντήσεις που γίνονται σε επίπεδο ε, εθνικών αξιωματούχων να μπορέσουν να λάβουν υπόψη αυτέ τι τροπολογίε. Στον επόμενο τριλόγο εμεί θα έχουμε μια παρουσίαση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να μα καταδείξει ποιε είναι οι τροπολογίε αυτέ οι τροποποίησεις οι οποίε μπορούν να γίνουν δεκτέ από τα δύο νομοθετικά θεσμικά όργανα. Έχουμε λοιπόν τις τροποποίησεις από το Κοινοβούλιο, έχουμε τις τροποποίησεις του Συμβουλίου, αλλά Υπάρχει μια συμφωνία γενικά ότι εμείς ως Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα τελευταίο σημείο, θα ήθελα να τονίσω και αυτό το σημείο, εμείς δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί η έννοια των διαδρόμων και ο ρόλος του συντονιστή για τα θέματα αυτά και εμείς θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη να παραμείνουν οι περιφερειακές περιοχές μέσα στα πλαίσια των διαδρόμων και αυτό θα έχει την, τις απαραίτητες επιπτώσεις για να χρηματοδοτηθούν και αυτές οι περιφερειακές περιοχές. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε την διατροπική διάσταση και την διαμεθοριακή διάσταση όλων αυτών των προγραμμάτων και όλα αυτά που αναφέραμε για την συμμετοχή των τοπικών αρχών, την δομή ε, σε διαδρόμους και όλα αυτά παραμένουν πάγια μας. Και όπως ανέφερε και ο κύριος ε, Κουμουτσάκος, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε με θεματικές ενότητες όλα αυτά τα θέματα και όχι να έχουμε χιλιάδες τροπολογίες. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε επί τη βάση θεματικών ενότητων στα θέματα αυτά. Κύριε Ρίκε, μια ερώτηση έχετε? Ναι. Ευχαριστώ τους εισηγητές. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση γιατί αρχίζουμε και τον τριμερή διάλογο για το ΣΕΕΦ. Και θα ήθελα να πω ότι ορισμοί ανάμεσα σε αυτό και τις κατευθυντήριες γραμμές έχουν συζητηθεί μεταξύ μας στο Κοινοβούλιο και έχουμε δεχτεί τους ίδιους ορισμούς για να υπάρχει συνοχή. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει συζήτηση στο Συμβούλιο για να αλλάξουν ή στις πρώτες διατάξεις της δεύτερης κάποιοι ορισμοί. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε ότι το Connecting Europe Facility με αυτό που εξετάζουμε τώρα πρέπει να διέπονται από συνοχή. Να είμαστε σαφείς λοιπόν με τους ορισμούς που έχουμε ήδη εγκρίνει, διότι αν αλλάξουν από τη μία από την άλλη μεριά, χαλάει η συνοχή και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργείται τότε. Γι' αυτό και προτείνουμε να μην αλλάξουν οι ορισμοί πάνω στους οποίους έχει συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δύο αυτά θέματα. Συστήνω λοιπόν στους συναδέλφους να φροντίσουν να κάνουν το ίδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές για να μην έχουμε πρόβλημα στο τέλος. Καλώς σχόλια. Γιώργο. Την παρέμβαση του Ντομινίκ και έχουμε ήδη διαμηνήσει και στην Προεδρία και στην Επιτροπή ότι θα είμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους του ΣΕΦ ανάλογα με τον βαθμό αλλαγών που μπορεί να γίνουν στους ορισμούς ακριβώς ό,τι είπε ο Ντομινίκ είναι και η δική μας θέση. Πρέπει να, πρώτα να συντονιστούμε μεταξύ ΣΕΦ και guidelines για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση και στον τρίλογο. Είναι δεδομένο, είναι αρχή μας, συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Can I now move on to the tachograph uh, one? This is the... Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, ποιος. Η κυρία Βιλμπάου. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω, ένα μικρό σχόλιο. Η Ιρλανδική Προεδρία κράτησε πολύ καλή στάση. Και η θέση τελικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σαφής. Χάρη βέβαια στις προσπάθειες που έγιναν από πριν. Και συμμερίζομαι επίσης το γεγονός ότι είναι θετικό το ότι δέχτηκαν τη μεθοδολογία. Ήταν το πιο προβληματικό οι έννοιες. Τώρα βέβαια πρέπει ακόμα να γίνει δουλειά για να έχουμε αυτή την προστιθέμενη αξία και συμμερίζομαι με τους εισηγητές τα όσα είπαν. Είμαι θετική απέναντι στην έκθεση αυτή, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντω πρέπει να μείνει στη στάση του όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, τη μεθοδολογία και κυρίως το ρόλο που παίζουν οι συντονιστές. Γιατί η έγκριση του κειμένου αυτού βέβαια είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να καθορίσουμε τις αρμοδιότητες των ατόμων εκείνων οι οποίοι δεν πρέπει να είναι ε, εργαλεία απλώς του διαλόγου, αλλά πρέπει να ευνοήσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τώρα το σχόλιο του κυρίου Έρτοκ για το πώς πάνε οι πολιτείς δημοσιονομικές προοπτικές. Εδώ πρέπει βέβαια να βάλουμε κάποια ποσά τα προγράμματα. Οι πολιτείς δημοσιονομικές προοπτικές, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν καλές. Οπότε ρωτάω, αν δεν το κάνουμε τώρα, μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε, να αναφερθούμε σε αυτά. Δεν συμφωνείτε. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Να το σκεφτούμε για το μέλλον. Επόμενο θέμα, ταχογράφη. Ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει ξανά και ξανά. Πρέπει να καταλήξουμε όμως κάπου. Παρακαλώ κύριε Τικάου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, συνεισηγητές μου. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω όμως τη γραμματεία της Επιτροπής μας για την ε, προσήλωσή τους και την υποστήριξή τους σε όλη τη διαδικασία διαδικασίας διαπραγματεύσεων για τα θέματα αυτά. Είχαμε πολλούς τριμερείς διαλόγους με την Κυπριακή Προεδρία. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν είχαν ακόμα επιτύχει μια πολιτική εντολή διαπραγμάτευση από το Συμβούλιο τότε. Ξεκινήσαμε πάλι τον τριμερή διάλογο με την Ιρλανδική Προεδρία. Έχουμε κάνει δύο άτυπες τεχνικού χαρακτήρα συναντήσεις ήδη. Και ο τρίτο. Ο δεύτερος μάλλον ε, τριγωνικός δίλογος γίνεται αύριο. Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η Ιρλανδική Προεδρία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να πείσει τα κράτη-μέλη και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά αμφιλεγόμενο στο Συμβουλίο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει τεχνικό χαρακτήρα, αλλά έχει και πολιτικές πτυχές. Αλλά η Ελλανδική Προεδρία έχει πραγματικά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα προκύψει ένα κείμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση συμφωνίας. Έχουμε λοιπόν καταγράψει κάποια πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο, έχουμε βελτιώσει την προστασία των δεδομένων, τις πρόνοιες για την προστασία των δεδομένων, έχουμε επίσης προχωρήσει σε συζητήσεις για την ε, τα στοιχεία που καταγράφονται στον ε, ταχογράφο και επίσης θα πρέπει να δούμε τις ε, διατάξεις για την αναβάθμιση των ε, οργάνων αυτών όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Γκρός. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την κατάσταση στους εθνικούς στόλους οχημάτων, φορτηγών οχημάτων. Επίσης έχουμε επίσης ε, προχωρήσει και στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα συνεργεία και τους ψηφιακούς ταχογράφους. Για τις κοινωνικές τώρα διατάξεις δυστυχώς εδώ το Συμβούλιο δεν έδειξε να θέλει να συζητήσει τα ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής νομοθεσίας. Για το Κοινοβούλιο όμως αυτά είναι εξόχως σημαντικά και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύουμε ότι η εξαίρεση για άτομα τα οποία, για οδηγούς οι οποίοι δεν οδηγούν επαγγελματικά, αυτό θα πρέπει να παραμείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μας ενδιέφερε. Θα προσπαθήσουμε θα προσπαθήσουμε, όπως είπα και πριν, να συζητήσουμε τα κοινωνικά θέματα, θέματα κοινωνικής νομοθεσίας με το Συμβούλιο, για τις κυρώσεις και την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Το Συμβούλιο δεν θέλει να προχωρήσει σε εναρμόνιση των κυρώσεων σε καμία περίπτωση. Ξέρω λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και θα χρειαστεί να έχουμε μια πιο εύκαμπτη θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο σημείο συζήτησης είναι τα θέματα κατάρτισης και η πιστοποίηση των ελεγκτών. Για την κατάρτιση, ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, για την πιστοποίηση το Συμβούλιο δεν θέλει να εφαρμόσει, να επιβάλλει κάποια μορφή πιστοποίησης η οποία θα κοστίζει πολύ και θα είναι πολύ κρατική κατά τη δική άποψη και εκεί το Κοινοβούλιο ίσως θα πρέπει να καταδείξει μεγαλύτερη ευελιξία. Υπάρχουν όμως σημεία όπου πρέπει να είμαστε αμετακίνητοι. Είναι ο εξοπλισμός ελέγχου. Και αυτό για ένα απλό λόγο. Το κύριο όφελος το οποίο προκύπτει από τη χρήση των ψηφιακών ταχογράφων είναι το γεγονός ότι θα έχουμε λιγότερους ελέγχους φορτηγών δεν θα σταματάμε τους οδηγούς που σέβονται την νομοθεσία, θα υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχων, επομένως θα σταματάμε μονάχα και θα ελέγχουμε τους οδηγούς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάποια όρια. Πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ελεκτικού μηχανισμού που γίνεται εξ αποστάσεως. Αν όμως δεν το κάνουμε αυτό, χάνουμε το όφελος. Απλώς θα έχουν όλοι οι μεταφορείς επενδύσεις, σε εξοπλισμό, σε κατάρτιση των οδηγών και τα συνεργεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτού του νέου εξοπλισμού. Εάν δεν υπάρχει μία ελάχιστη χρήση ελεγκτικού εξοπλισμού, εμείς δεν μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτές τις ε, πρόνοιες. Για το Κοινοβούλιο λοιπόν ο εξοπλισμός ελέγχου παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαστε ευέλικτοι για την ε, τροποποίηση του κειμένου μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, παραδείγματο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε το κείμενο του Συμβουλίου με την τωρινή μορφή που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μην χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εξοπλισμό. Αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο για μας και είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πραγματικά ανεπαρκές ως μήνυμα προς τους μεταφορείς ότι λόγω της κρίσης μπορούν να εξαιρεθούν από όλα αυτά τα μέτρα. Και τέλος, οι εφαρμοστικές πράξεις, η, η κατεξουσιοδότηση πράξη. Εμείς είχαμε την εντολή να υποστήριξουμε τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Το, το Συμβούλιο όμως θέλει εφαρμοστικές πράξεις και θέλει να αφαιρέσει και το παρατημα ένα 1β θέσαμε το ερώτημα στις νομικές υπηρεσίες των δύο θεσμικών οργάνων με την υποστήριξη της Κομισιόν για να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο νομικών υπηρεσιών και έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που είναι ικανοποιητικό για όλους. Ίσως θα χρειαστεί να δείξουμε εδώ κάποια ευελιξία ώστε να καταλήξουμε σε μια περιορισμένη αλλά σαφή εντολή για την Κομισιόν, είτε πρόκειται για εφαρμοστικέ είτε κάτι εξουσιοδότηση πράξη. Αλλά θα πρέπει να περιορίσουμε αυτή την εντολή που δίνουμε στην Κομισιόν. Γι' αυτό το λόγο εισαγάγαμε στο κύριο κείμενο ορισμένε τροπολογίε. Και σήμερα οι νομικές υπηρεσίες θα συναντηθούν. Ελπίζω ότι θα προκύψει κάτι και αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο θεσμικών οργάνων. Ελπίζω ότι αύριο στον τριμερή διάλογο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα 95% των πολιτικών πολιτικού χαρακτήρα θεμάτων και κατά τη διάρκεια της Ιλλανδικής Προεδρίας ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και τα 5% που παραμένει. Για την άποψή μου είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συμφωνία μέσα στην διάρκεια τη Ελληνική Προεδρία, γιατί έχουν καταβάλει τεράστιε προσπάθειε που τι αναγνωρίζουμε. Θα ακολουθήσει η Λιθουανική Προεδρία και μετά η Ελληνική Προεδρία και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι λιγότερο διαθέσιμοι για να συνεργαστούν μαζί μα για το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την, μέσα στην ελληνική Προεδρία. Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις. Θα ήταν ε, σύντομε παρουσιάσει των αποτελεσμάτων των τριμερών διαλόγων, είχαμε πει στην αρχή, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω πραγματικά να είμαι σύντομη. Καταρχήν ευχαριστώ τη Σίλβια. Ήταν πολύ σκληρέ οι διαπραγματεύσει και είναι αλήθεια πρέπει να κλείσουμε τώρα στην Ιρλανδική Προεδρία, αλλιώ τα πράγματα είναι πολύ μαύρα. Και δύο πράγματα η μετασκευή του ταχογράφου. Αυτό ε, πράγματι το πείραγμα όπως λέμε ε, μπορεί να ισχύει μόνο για τις ε, διεθνείς διαδρομές. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε τα 100 χιλιόμετρα όπως ε, προτείνονται να είναι ο κανόνας και όχι η εξέρεξη και επίσης και τα αμαξίδια, αμαξάκια των εργοταξίων ε, και αυτά κάπως πρέπει να τα εξετάσουμε. Το Συμβούλιο λέει ότι δεν θέλει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δείξουμε και εμείς καλή θέληση αν θέλουμε σε άλλα θέματα να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες του Συμβουλίου. Ωραία, το Συμβούλιο ξέρω ότι είναι λιγάκι σε πανικό με όλα αυτά τα θέματα. Το στοιχείο κλειδί είναι ότι και εμείς πρέπει να είμαστε ελαστικοί. Αυτό να έχουμε υπόψη μας. Παρακαλώ κύριε Γρός. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομο. Ο συνάδελφο ε, κύριο Χεγγίνης ε, έπρεπε να φύγει και θέλω να, επέμβω, να παρέμβω σε δύο-τρία θέματα και να πω ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε την οικονομία αν δεν τιμωρήσουμε την μεσαία τάξη, για να το πω έτσι απλά. Και στο Κοινοβούλιο κάναμε την πρόταση, αντί να έχουμε 20 ε, σελίδε εξαιρέσει, απλά τους μη επαγγελματίες να τους εξαιρέσουμε από αυτή την οδηγία. Ε, πώς, ας πούμε, μπορώ να εξηγήσω στον ε, σκεπά μου αυτό που μου κάνει τη σκεπή ότι όταν τελειώσει τη δουλειά του δεν μπορεί να γυρίσει το βράδυ σπίτι του. Επίσης, αυτά που πολλοί φαντάζονται αυτή τη στιγμή θα χαθούν για ολόκληρη την Ευρώπη. Και όσον αφορά το ε, αποτέλεσμα ως διατυπώνεται δεν θα οδηγήσει πουθενά. Είτε θα το δεχτούμε αυτό που λέμε, είτε αύριο θα είμαστε αναγκασμένοι να αγοράσουμε κινέζικα και ρωσικά μοντέλα. Αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε στους πολίτες. Ε, εμείς από πλευράς ΕΛΚ θέλω να σας πω ότι αν δεν επιτυγχάνεται η προστιθέμενη αξία, δεν θα δεχτούμε την πίεση του χρόνου που ασκείται και δεν ε, θα δεχτούμε και το αποτέλεσμα. Ωραία, είπαμε. ότι αυτές θα ήταν παρουσιάσεις συμπερασμάτων από τις ε, συνδιαλλαγές. Μην ε, μπαίνουμε τώρα στην ουσία του θέματος για το σταχογράφους. Ίσως κακός ήμουν τόσο γενναιόδωρος και είπα ότι μπορούμε να έχουμε εδώ αυτές τις παρουσιάσεις. Συνήθως θα κάνουμε μεταξύ συντονιστών. Τέλος πάντων, ο κύριος Αλκαντροή. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να αντιδράσω λίγο σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπρος πριν από λίγο. Και εγώ είμαι υπέρ τη ελαστικότητα, αλλά προσοχή, γιατί είναι δύσκολο να φτιάξουμε τους ορισμούς προσθέτοντας εξαιρέσεις. Πρόεδρος, κύριε Αλκαδραουή, γνωρίζετε ότι έχουμε μία εντολή. Το μόνο το οποίο διαπραγματευόμαστε δεν είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής και πάνω σε αυτήν βασιζόμαστε για τις διαπραγματεύσεις. Καλώς, εγώ θέλω απλώ να το επιβεβαιώσουμε αυτό για να μην αρχίσει πάλι η συζήτηση αυτή από πλευράς της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου, λέει ο κύριος Σελκαντρουή. Πρόεδρος, καλώς. Ωραία, τότε Υπενθυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα αρχίζουμε στις 3 και μισή, όχι στις 3, 3 και μισή. Οπότε μετά από αυτή τη μεγάλη ψηφοφορία που είχαμε, έχετε και μισή ώρα παραπάνω διάλειμμα.